Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Προτείνω να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Να συνεχίσουμε τις επαφές που έχουμε με τη Σουηδική Προεδρία εχθές. Κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή με μία από τις συναδέλφους σας. Κύριε Σβέν Ότο Λιτορίν, θα συνεχίσουμε με εσά σήμερα. Είστε Υπουργό Εργασία και άρα προεδρεύετε στο Συμβούλιο Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι μεγάλη μα τιμή που σα υποδεχόμαστε σήμερα στην Επιτροπή μα. Δυστυχώ η συνάδελφό σα, η Χριστίνα Χιούσμαρκ Πέρσον, που είναι αρμόδια για την κοινωνική ασφάλιση, χρειάζεται και σήμερα την κοινωνική ασφάλιση γιατί έπαθε μια γρήπη. Δεν λέω πια γρήπη τώρα, αλλά... Αλλά ε, ε, η υφυπουργός Μπετίνα Σπιπή την αντικαθιστά Λοιπόν, προτείνω να κάνετε εσείς τις ε, παρουσιάσεις σας για το πρόγραμμα τη Προεδρίας και μετά κάνουμε τι ε, τις ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να ε, ζητήσω συγγνώμη από τη συνάδελφό μου που δεν μπορούσε να έρθει. Δεν ε, ε, έχει την γρήπη των χείρων ή όπως και να τη λέμε αυτή τη γρήπη. Απλώς είναι άρρωστη. Θα ήθελα να προσπαθεί σήμερα να σας μιλήσω αγγλικά. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν τα σουηδικά, αλλά ίσως Τα αγγλικά είναι μια κοινή γλώσσα και υπάρχουν κοινοί όροι, αν θέλετε, ε, κατανοητοί από όλου μα. Γαλλικά θα και τα γαλλικά ίσως είναι το ίδιο διαδεδομένα εδώ, αλλά δεν ε, ε, νομίζω ότι τα καταφέρνω καλά σε αυτή τη γλώσσα. Αν πάση περιπτώσει, χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα ήθελα να σας πω μερικά πράγματα για το πρόγραμμα εργασίας της Σουηδικής Προεδρίας. Όπως φαντάζεστε όλοι, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αν θέλετε της Σουηδικής ε, Προεδρίας επηρεάστηκε σημαντικά από τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία ε, διατρέχει η Ευρώ... και η Ευρώπη μια οικονομική κρίση. Τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία και συγχρόνως υπάρχουν βεβαίως και κάποια βασικά σημεία που ε, παραμένουν σταθερά. Έχουμε πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους εκτός αγοράς εργασίας. Βεβαίως μεγάλη ανεργία υπήρχε και πριν από την κρίση. Απλώς η κρίση επιδεινώνει τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα ε, εκεί ε, τα οποία δεν επηρεάστηκαν από την διεθνή κρίση αλλά δημιουργούν ανησυχίες. Η κρίση ωστόσο δεν είχε απροσδόκητα και προφανώς αρνητικότατα ε, αποτελέσματα, επιπτώσεις στις αγορές εργασίας. Ε, μερικοί μιλούν τώρα για την κρίση που έχει σχεδόν περάσει και ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες απαρχές βελτίωσης. Δεν θέλω εγώ να παίξω το μάγο εδώ και να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις. Ε, Εκείνο που θέλω να κάνω είναι να φέρω κάποια σημαντικότατα ε, θέματα τα οποία κατά την άποψή μου αξίζει να συζητηθούν και ε, μέτρα να παρθούν σχετικά τους επόμενους μήνες. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι τελικά η κρίση θα τελειώσει κάποια στιγμή. Ιστορικά υπήρχαν ε, στο παρελθόν και άλλες οικονομικές κρίσεις θυμηθείτε την κρίση της τουλίπας της Ολλανδικής το 1637 υπήρχαν πολλές λοιπόν οικονομικές κρίσεις ε, τις οποίες, ε, ε, από τις οποίες επιβιώσαμε έξι οικονομικές κρίσεις θα μπορούσε να μετρήσει κανείς στο παρελθόν τούτη εδώ είναι η έβδομη που βιώνουμε αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακόμη σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία γίνονται προφανείς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αγορές εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και εκείνο που θέλουμε εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να προλάβουμε και να δράσουμε τόσο ώστε να μην παραμείνουμε στα επίπεδα ανεργίας τα οποία αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά. Η πείρα μας λέει ότι τα άτομα τα οποία δεν εργάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ε, κινδυνεύουν να βρεθούν μονίμως αποκλεισμένα. Άρα πρέπει να είμαστε ενεργοί, πρέπει να παρεύουμε έγκαιρα, να εφαρμόσουμε μέτρα ε, στην εκπαίδευση, να προσπαθήσουμε να ε, προλάβουμε ορισμένα πράγματα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως ε, υπάρχουν μέτρα συντονισμένα τα οποία πάρθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ε, σχεδίου ανασυγκρότησης και που βοηθούν την κατάσταση. Ε, υπάρχουν όμως και άλλα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε. Παραδείγματο χάρη υπάρχει το θέμα της μικροοικονομικής, μικροδανείων, μικροπιστώσεων κτλ. Η σχετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, δίνουμε μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό και ελπίζουμε να και ήδη ξεκίνησαν οι σχετικές συζητήσεις και πραγματικά πιστεύουμε να συνεχιστούν και να πάρθουν αποφάσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γιατί πιστεύουμε ότι το μέτρο αυτό μπορεί να βοηθήσει πραγματικά θα ήταν πολύ σημαντικό επίσης μήνυμα προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να ξεκινήσουν και κάποιες άλλες ε, δράσεις ε, στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη. Βεβαίως, η, ε, στόχος μας ήταν ανέκαθεν και είναι ακόμη περισσότερο τώρα να δημιουργήσουμε αγορές εργασίας στην Ευρώπη βιώσιμες. Όλοι φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι η απασχόληση, εργασία είναι βασικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και για τα μεμονωμένα άτομα και για την κοινωνία στο σύνολό της. Δεν μπορεί η Ευρώπη να υστερήσει στο, ή να αδρανήσει σχετικά με θέματα απασχόλησης. Πιστεύουμε ότι ε, όλοι πρέπει να είναι μέρος, έχουν δικαίωμα να είναι μέρος της αγοράς εργασίας και ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Θέλουμε να μην έχουμε πολίτες που απλώς παίρνουν τα επιδόματα της κοινωνικής ασφάλισης. Θέλουμε να γίνουν φορολογούμενοι άνθρωποι αυτοί, να βρουν δουλειά, να δουλέψουν, να γίνουν φορολογούμενοι. Αυτό είναι η προστιθέμενη αξία πέραν του ότι οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν δουλειά. Θέλουμε λοιπόν να ενδυναμώσουμε τα θεμέλια των αγορών εργασίας στην Ευρώπη και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κατά την άποψή μου μια Ευρώπη με κοινωνικό πρόσωπο ξεκινάει από τις θέσεις εργασίας Λοιπόν, θέλουμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι οι δημογραφικές τάσεις, η δημογραφική πρόκληση είναι πρόβλημα, δεν πρόκειται να αλλάξει όμως. Ε, θέλουμε λοιπόν βιώσιμη ανάπτυξη, ευημερία ε, στην κοινωνία μας Θέλουμε όσο δυνατόν περισσότεροι από τους πολίτες μας να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και βεβαίως είναι εύκολο να το λέμε αυτό, ε, αλλά ε, και τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη ανάλογα με ιστορικές αν θέλετε και πολιτικές ε, ε συνιστώσεις. Πιστεύουμε όμως ότι ο στόχος όλων πρέπει να είναι για την Ευρώπη ε, υγιή οικονομία, υγιείς αγορές εργασίες ε, και υγιής απασχόληση, μικρή ανεργία. Βεβαίω αν θέλουμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, να αντιμετωπίσουμε επίσης την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει η... μέσα να βάλουμε τα ζητήματα αυτά με υψηλή προτεραιότητα μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας. Τον Ιούλιο στην άτυπη Υπουργική Σύνοδο του Γιον Κόπινγκ ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για τα θέματα αυτά οι οποίες θα συνεχιστούν και θα προωθηθούν τώρα το φθινόπωρο και η Προεδρία πιστεύει ότι πρέπει να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στις συζητήσεις αυτές. Ε, θέλω να ε, έχω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την ε, Επιτροπή σας και η επόμενη ευκαιρία να συζητηθούν τα θέματα αυτά θα είναι το, η συνδιάσκεψη ψηλού επίπεδου που θα γίνει στη Στοκχόλμη το τέλος, στο τέλος Οκτωβρίου θεωρούμε ότι είναι αδύρυτη η ανάγκη να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν αγορές εργασίας πιο ενισχυμένες ε, και πιο συνεκτικές και αυτός είναι ο στόχος, αυτό το στόχο θα προωθήσουμε τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Και εγώ ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Ε, χωρίς ε, καθυστέρηση θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπετίνα Κασιφή. Έχετε το λόγο παρακαλώ κυρία μου. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω σου ειδικά, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω και πάλι ότι η Κριστίνα Χιούς Πέρσον ε, λυπάται πάρα πολύ που δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση γιατί ήθελε πάρα πολύ να σας συναντήσει και να παρουσιάσει το πρόγραμμά της σήμερα. Τι να κάνουμε, πάντως είναι τιμή για μένα που έχω εγώ την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα ζητήματα που έχει αναδείξει προτεραιότητα η Υπουργός μας ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας αρχικά. Θα ήθελα να επανέλθω στο εξή ζήτημα. Πόσο μπορούμε να έχουμε μια αγορά εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου θα συμμετάσχει ένα μέγιστο αριθμό ε, ατόμων, όπω μα είπε ο Υπουργό Βενότο Λιτορίν στην πρώτη παρουσίαση. Είναι καταλητικού χαρακτήρα αυτή η ερώτηση, ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε τον αποκλεισμό που βιώνουν πολλοί άνθρωποι σήμερα για να δημιουργήσουμε τέτοιες αγορές εργασίας ε, όπου συμμετέχουν ε, οι περισσότεροι άνθρωποι, χρειάζεται μια στενή σχέση ανάμεσα στην ε, πολιτική απασχόλησης και την πολιτική κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή στενή συνεργασία ανάμεσα στον Υπουργό Απασχόλησης και στο, στην Υπουργό Αρμόδια για την κοινωνική ασφάλιση. Από κοινού φέρνουν την ευθύνη για να προάγουν αυτή τη προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και εν του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ και γι' αυτό ήρθαμε να σας συναντήσουμε σήμερα. Προς το παρόν διερχόμεθα μια πολύ δύσκολη περίοδο οικονομικής κρίσης και όπως είπε ο υπουργό Λιτορίνε είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι είναι προσωρινή αυτή η κρίση και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που αναλαμβάνουμε λόγω αυτής της κρίσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους μακρόπνους ε, στόχους μας ε, για να δημιουργήσουμε αυξημένη απασχόληση και μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Δεν ε, επιτρέπεται όσοι είναι σε ηλικία να εργαστούν και λόγω της κρίσης ε, ζουν από τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να τους να επιτρέψουμε να παραμείνουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ε, αέργοι και αποκλεισμένοι. Συγγνώμη. Αυτό είναι βασικό ζήτημα για το κράτος πρόνοιας και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Ο στόχος μας είναι να, να έχουμε μια βιώσιμη κοινωνία, βιώσιμη από οικονομική και από κοινωνική άποψη. Το φθινόπερο θα γίνει μια συζήτηση σχετικά με το πώς με τη βοήθεια μιας ενεργούς πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης σε συνεργασία με μια ενεργή ε, πολιτική απασχόλησης ε, για μέγιστη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού. Πώς λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλους. Ε, μια τέτοια πολιτική δίνει υποστήριξη και κίνητρα για δουλειά για όσους ε, δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας για λόγου υγείας. Ε, σε αυτή την πολιτική εντάσσονται και προληπτικά μέτρα για να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων, δηλαδή την αποχή από την αγορά εργασίας για λόγους υγείας. Μια ενεργός πολιτική κοινωνικής ασφάλισης δημιουργεί τέτοιε προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι βάσει των δυνατοτήτων τους ε, εισέρχονται στην αγορά εργασίας και μια τέτοια πολιτική δεν ευνοεί μόνο όσους καλύπτονται από το σύστημα απασχόληση και από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει, και όσους έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την αγορά εργασίας και δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν και να νιώσουν ότι συμμετάσχουν στην κοινωνία ε, και άρα προβάλλουμε το ρόλο των ατόμων μέσα στην κοινωνία. Στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Γεν Σόπινγκ που έγινε τον Ιούλιο, αρχίσαμε μία συζήτηση σχετικά με το πώς θα δημιουργήσουμε αυτές ε, τις ε, αγορές εργασίας όπου εντάσσονται οι περισσότεροι άνθρωποι της κοινωνίας και είχαμε πάρα πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και υπήρξε ευρεία υποστήριξη για την συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με την ενεργό πολιτική κοινωνικής στο φθινόπωρο. Ε, στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τις αγορές εργασίας ε, που προανέφερε και ο Υπουργό Λειτουργών, που θα λάβει χώρα στη Στοκχόλμη στις 26 και 27 Οκτωβρίου. Στη διάσκεψη αυτή, οι πολιτικοί, οι εμπειρογνώμονες και οι εκπρόσωποι διαφόρων οργανώσεων πρόκειται να συνεχίσουν αυτή την συζήτηση και ο στόχος είναι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας να οδηγήσει η συζήτηση αυτή σε ένα σαφέ μήνυμα από το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ε, και να αποδοθεί νέο περιεχόμενο στη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση που θα εγκριθεί την ερχόμενη άνοιξη υπό Ισπανικής Προεδρίας. Ε, η υλοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ε, εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης ζωτική σημασία για την απασχόληση επίπεδο Ένωσης. Μετά από δουλειά πολλών ετών, εσχάτως καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ένα νέο εκμοντενισμένο και απλουστευμένο νομικό πλαίσιο, ώστε να συντονίσουμε τα ε, συστήματα κοινωνικής ασφάλειας των κρατών μελών. Αυτό το νομικό πλαίσιο ε, είναι μία εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση ούτως ώστε να έρχονται οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να μετακινούνται μάλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε να εργαστούν ή να σπουδάσουν σε μία άλλη χώρα. Και ε, με πάσα νομική ασφάλεια βλέπουμε ότι ε, λειτουργούν αισίως αυτοί οι κανόνες περί συντονισμού και είμαι Χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά υπήρξε συνένεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή σε όλες τις προηγούμενες προεδρίες που συνεισέφεραν στην έγκριση του κανονισμού 883 04 και τον εκτελεστικό του κανονισμό μετά από ε, δεκαετή εντατική εργασία και τελικά μπορεί πλέον να τεθεί σε ισχύ την 1η Μαΐου του 2010. Ο νέος ε, κανονισμός συνεπάγεται ε, σημαντικές ευελτιώσεις. Οι δημόσιες διοικήσεις απλουστεύονται και γίνονται πιο αποτελεσματικές και η ασφάλεια δικαιού για τους πολίτες της Ένωσης αυξάνεται. Ένα σημαντικό καθήκον για μας το φθινόπωρο είναι να προετοιμάσουμε και τους πολίτες και τα κράτη-μέλη και τις διοικήσεις κοινωνικής ασφάλισης, αρχές κοινωνικής ασφάλισης, ε, ούτως ώστε να εφαρμοστούν οι νέες αρχές. Πρέπει να εργαστούμε εντατικά, ούτως ώστε να υπάρξει και καλή συνεργασία ανάμεσα σε εθνικές αρχές. Το φθινόπωρο θα οργανώσουμε διάφορα σεμινάρια για θέματα κοινωνικής ασφάλισης και η έκβαση των σεμιναρίων, τα πορίσματα θα ομαδοποιηθούν σε μια διάσκεψη που οργανώνουμε την Στοκχόλμη από τις 25 ως τις 27 Νοεμβρίου του 2009. Ένα σημαντικό ζήτημα για το συντονισμό των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών ως προς αυτούς τους κανόνες και υπάρχει και σχετικός κανονισμός. Ε, οι υπήκοοι τρίτων χωρών ε, έχουν δικαίωμα, τα ίδια δικαιώματα όπως και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το που μετακομίζουν και εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση τα ίδια δικαιώματα ως προς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Απαραίτητος πρέπει να προσαρμόσουμε τους εθνικούς κανόνες τον νέο κανονισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αναβαθμιστεί η προστασία ως προς την κοινωνική ασφάλιση των υπηκών των τρίτων χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνεπάγεται επίσης διοικητικές απλουστεύσεις διότι θα εφαρμόζονται πολύ απλά ενιαίοι ομοιόμορφοι κανόνες για όλους ανεξαρτήτως ε, υπηκότητας και παρά τις εντατικές προσπάθειες της Τσεχικής Προεδρίας οι Υπουργοί στις 9 Ιουνίου στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ε, για ένα νέο κανονισμό για την προσαρμογή των κανόνων συντονισμού ως προς τους υπηκούς των τρίτων χωρών. Η δική μας Προεδρία θα συνεχίσει να προσπαθεί ούτω ώστε να βρούμε μια λύση ε, που θα μπορέσουν να δεχτούν όλα τα κράτη-μέλη η οποία λύση όμως δεν θα συνεπάγεται επιδείνωση κατάσταση των επικών τρίτων χωρών σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Περιμένουμε με ανυπομονησία την ενδιαφέρουσα και επικοδομητική συζήτηση που θα γίνει σήμερα στην Επιτροπή σας για τις εργασίες του Φθινόπορου. Ευχαριστούμε. Merci Ευχαριστούμε. Έχουμε λίγο παραπάνω από μία ώρα για την ε, συζήτησή μας. Έχουμε ήδη 10 ομιλητές στον κατάλογο. Je les prends dans, dans l'ordre de... Ας ε, τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, με τη σειρά εγγραφή στον κατάλογο. Ροβάνα Πλόμπ και Ρίχαρτ Φάλμπ μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους υπουργούς στην Επιτροπή μας και στον ε, πρόεδρο του Συμβουλ... Ε, που προεδρεύουν του Συμβουλίου. Με ικανοποίησαν ιδιαίτερα οι πληροφορίες και θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Dacă vor folosi în pregătirile pentru anul 2000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 μας ενδιαφέρει τι θα γίνει το 2010 που θα έχουμε θέματα ε, κοινωνικού αποκλεισμού και θα είναι το χρώμα για, ε, ε Ευρωπαϊκό για την Ένδια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Υπάρχουν πράγματα, τα ε, άτομα τα οποία είναι εκτός αγοράς εργασίας, υπάρχουν διακρίσεις για τους νέους και τις γυναίκες και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό και θα πρέπει να προβλέψουμε ένα σχέδιο δράσης για να, να μειωθεί αυτό το κενό και στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας. Έχετε πρόθε, προτίθεστε η τη στρατηγική αυτή που αποφασίστηκε το 2008 για τον κοινωνικό αποκλεισμό να την εφαρμόσετε εκεί προβλέπεται και ένας ελάχιστος μισθός ο οποίος είναι κατά την άποψή μου πολύ σημαντικός διότι εξασφαλίζει μια ελάχιστη αξιοπρέπεια στον πολίτη ακούσουμε τέσσερις ερωτήσεις, αυτό σας προτείνω και μετά να σας δώσουμε το λόγο για να μην διαφύγετε άμα ακούσουμε αμέτρητες ερωτήσεις. Ρισάρτ Φάλμπρ και η κυρία Ελίζαμπεθ Σρέντερ. Η Σουηδία είναι μια χώρα την οποία εμείς από τις νέες χώρες μέλη θεωρούμε ε, υπόδειγμα. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να σας πω ότι και οι δύο παρουσιάσεις των Υπουργών ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικές για μένα. Ε, δεν είπατε τίποτα για τα κοινωνικά προβλήματα. Τι γίνεται με την υπόθεση Λαβάλ, η οποία απειλεί τις θέσεις των συνδικάτων στις ε, ευρωπαϊκές χώρες. Η στρατηγική της Λισαβόνας Όπως είπε ο ε, Επίτροπος Σπίτλα, ο οποίος διακρίνεται για την έλλειψη χιούμορ του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ε, σημασία έχει το σχολείο του, είναι ένα γέτη, είναι ένα τέρας το οποίο δεν έχει δει κανένας ε, ποτέ. Αρχίζουμε και εννοούμε συνέχεια όρους, ε, flexicurity, το ένα, το άλλο. Πότε θα αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει η Ευρώπη. Και εδώ σας μιλάω για τη σταδιακή κατάρρευση του εργασιακού δικαίου και των διεθνών συμφωνιών του Διεθνούς Οργανισμού Εργασία ουσιαστικά τα συνδικάτα σιγά σιγά αποδυναμώνονται και εγώ περίμενα από εσά απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Άκουσα τους δύο υπουργού σήμερα και μου δόθηκε εντύπωση ότι ε, κάποια τσέχικοι γρήφοι έχουν πάθει, γιατί οι Τσέχοι δεν τα πρόσεξαν καθόλου αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το δύο εκπροσώπους της Σουηδικής Προεδρίας εδώ. Θα ήθελα εμπολής να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Φάρμπερ ε, διότι και εμεί θεωρούμε την Σουηδία πρότυπο στον τομέα τη απασχόληση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων. Αυτά δεν αναφέρθηκαν όμως καθόλου στις ομιλίες των Υπουργών. Ε, ε, ξέρουμε ότι ε, μάλλον γίνεται συζήτηση για το ότι κάποια δικαιώματα των γυναικών που ορίστηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο τελικά από μια απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει ίσως να ε, προστατευτούν περαιτέρω να αναθεωρηθεί η σχετική οδηγία. Αλλά εκείνο που με απασχολεί αλλά δεν ξέρουμε ποτέ αν θα γίνει αυτό στην Ευρώπη και δεν το ανέφερε και η Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα ε, όμως ε, να ρωτήσω πιο συγκεκριμένα τη Σουηδική Προεδρία για το τι θα κάνει με την οδηγία αυτή των αποσπάσεων ε, και το, τα δικαιώματα των ε, γυναικών. Επίσης ε, δεν άκουσα τίποτα δεν, δεν άκουσα τίποτα γενικά για πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Εντίθε Στρέλα τώρα στην προηγούμενη θετία ήταν η συγγήτριά μας για την οδηγία για τις ε, άδειες μητρότητας. Έχετε το λόγο, αλλά η κυρία Στρέλα μιλάει εκτός μικροφώνου και δεν την ακούμε εμείς. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους υπουργούς, να τους ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις τους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την οδηγία που είναι γνωστή για, ως ε, οδηγία άδειας μητρότητας. Ε, στην Επιτροπή Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων ήμουν εισηγήτρια για αυτή την οδηγία και στο Στρασβούργο ήδη έχω συναντήθηκα με τον ε, αξιότιμο Υπουργό. Έχουμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια έγινε μια πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή Γυναικών και είχαμε και άλλες επαφές ε, στο μεταξύ με την Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μου πείτε, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ζητήματος και λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες μας, ε, αυτές που έγιναν στην προηγούμενη θητεία και επίσης λαμβάνοντας υπόψη ε, την... το ότι είναι αυθεντία, αν θέλετε, η Σουηδία, γιατί είσαστε πολύ προοδευτικοί σε αυτό το τομέα. Θεωρείτε λοιπόν κύριε Υπουργέ πιθανό να προκύψει συμφωνία στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας ή να το πω απλά ποιες είναι οι προσδοκίες σας για αυτό το φάκελο. Um, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ εύστοχες και πολύ καλές οι ερωτήσεις σας ε, για όλα αυτά τα θέματα. Καταρχάς να σας πω κύριε Πλάμ ότι η συμπερίληψη των ομάδων που είναι λιγότερο ενεργές ε, στην ε, αγορά εργασίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που προσπαθούμε να διευθετήσουμε. Ο λόγος είναι φυσικά ε, Ας δούμε για παράδειγμα τους ανθρώπους που έχουν μια κάποια αναπηρία, έχουν προβλήματα στην αγορά εργασίας ε, και δεν είναι αποδεκτό αυτό, όχι μόνο για λόγους διακρίσεων, αλλά και για λόγους ευρύτερης κοινωνίας χρειαζόμαστε οποιονδήποτε μπορεί να δουλέψει στις αγορές εργασίας μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δημογραφικές προκλήσεις που μας περιμένουν, αλλά και ταυτόχρονα να συνδράμουμε στην παραγωγή για να μπορέσουμε να έχουμε σχολεία και πρόνοια ε, για το μέλλον. Τώρα, Βάσει των όσων μας επιτρέπουν οι συνθήκες, η στρατηγική μετά τη Λισαβόνα, μετά από το 2010, είναι το πλαίσιο στο οποίο θα θέλαμε να εστιάσουμε τις ενεργειές μας. Επιπλέον, θα πρέπει να επεξεργαστούμε κάποιες οδηγίες και κάποιες ε, κανονισμούς που μας ε, αφορούν και έχουν να κάνουν με τον τομέα της απασχόλησης αλλά θέλουμε επίσης να βρούμε και τα κατάλληλα κίνητρα για να ενταχθούν οι άνθρωποι στην αγορά εργασίας και να υπάρχουν ε, ταυτόχρονα και αποτρεπτικά ε, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να άρουμε, όπως για παράδειγμα τους χαμηλούς μισθούς, ε, τα μη ευνοϊκά συμβόλαια κλπ. Ο ελάχιστος κατώτατος μισθός είναι κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος για να είμαστε ειλικρινείς και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές εργασιακές συνθήκες θέλετε. Για παράδειγμα, εμείς στη Σουηδία δεν έχουμε καμία νομοθεσία για τη μισθοδοσία. Εμπιστευόμαστε τους κοινωνικούς εταίρους μας και πιστεύουμε ότι θα είναι υπεύθυνοι για την ε, διαδικασία ε, προσαρμογής των μισθών και δεν θα θέλαμε οι πολιτικοί να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία διαμόρφωσης των μισθών και για να είμαι ειλικρινής εμείς στη Σουηδία αυτό το σύστημα θα θέλαμε να διαθετηρήσουμε. Και παρά το γεγονός ότι κατανοώ ότι εσείς έρχεστε από μια διαφορετική χώρα και σας ενδιαφέρει το θέμα των των μισθών και της ίσης ε, των λιγότερων ευνοημένων, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο που βοηθούν, να βοηθήσουμε ανθρώπους που χρειάζονται συνδρομή για να ενταχθούν στην αγορά εργασία. Ε, το βασικό όμως είναι ότι χρειαζόμαστε τον οποιονδήποτε μπορεί να εργαστεί στην αγορά εργασίας για να μπορέσουν να λειτουργούμε τα συστήματα ασφάλισης μας στο μέλλον. Ελπίζω να απαντώ στην ερώτησή σας. Κύριε Φάλμπερ και η κυρία Σρέντερ, αναφερθήκατε στην υπόθεση Λαβάλ. Ε, έχω παραστεί και στο παρελθόν εδώ που συζητήσατε κάποια θέματα και κάποια θέματα για τις δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Δυστυχώς ε, το αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν μας ικανοποίησε. Όταν είδαμε τα αρχικά προκαταρκτικά αποτελέσματα θεωρήσαμε ότι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε την κατάσταση στην οποία έχουμε βρεθεί αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε το θέμα από δύο πρόπτικε. Το ένα έχει να κάνει με την εθνική μα νομοθεσία και το άλλο έχει να κάνει με το τι μπορεί να γίνει, τι θα πρέπει να γίνει ή θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που συνέβη είναι ότι μόλι λάβαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εγώ κάλεσα του κοινωνικού εταίρους στη Σουηδία και του ζήτησα να συμμετάσχουν σε μια γενική συζήτηση στη Σουηδία για το πώ θα αντιμετωπίσουμε ε, την ε, κατάσταση που προέκυψε. Επίσης ξεκίνησε και μία έρευνα για τη διαδικασία ε, και αυτή έγινε σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Η έρευνα αυτή ε, είχε ως αποτέλεσμα μία έκθεση. Αυτή την έκθεση αυτή τη στιγμή την εξετάζει η κυβέρνηση και σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε σχέδιο νόμου στο Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση σε εσωτερικό επίπεδο. Εσωτερικός καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν περίπου 2 ε, με 3.000 χιλιάδες αποσπασμένοι εργαζόμενοι στο, ε, στη Σουηδία. Οι περισσότεροι από αυτούς καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις της Σουηδίας, επομένως μιλάμε για μερικές εκατοντάδες ανθρώπους. Αυτό βέβαια στην πράξη μπορεί να μην είναι μεγάλο, αλλά από ε, νομική σκοπιά εξακολουθεί να είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, αν θέλετε να δείτε περισσότερα πράγματα, στην ε, ε, ιστοσελίδα της κυβέρνησή μας υπάρχει μία σύνοψη στην αγγλική και θα μπορούσαμε να σας δώσουμε και περισσότερες ε, πληροφορίες για το πώς αντιμετωπίζουμε εσωτερικό στην κατάσταση. Είμαι βέβαιος ότι μέσω της νομοθεσίας που θα παρουσιάσουμε στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με όσο το δυνατόν πιο λογικό τρόπο. Και θα έχουμε διαφυλάξει το σουηδικό μοντέλο όπως ε, θα θέλαμε να παραμείνει. Βέβαια, η δική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε και συλλογικέ συμβάσεις αλλά και συλλογικέ δράσεις ε, αν παραστεί ανάγκη στην αγορά εργασίας μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ακαθόδη για να είμαι ειλικρινής. Άκουσα δύο ερωτήσεις και δύο πιθανές απόψεις. Η μία ήταν να αλλάξει η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους και το άλλο θα ήταν να αλλάξει η συνθήκη και να συμπεριλάβει κάτι για το θέμα. Αν ε, έχουμε μια κοινωνική ρήτρα ε, στην ε, συνθήκη, αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό βήμα και αυτό είναι και ο λόγος για του οποίου εγώ προασπίζομαι την κύρωση της συνθήκης ε, που σημαίνει ότι θα τεθεί σε εφαρμογή γιατί κατά την άποψή μου αυτό θα είναι λύση του προβλήματος. Η κοινωνική ρήτρα βέβαια θα πρέπει να κατανοήσω πρώτα τι σημαίνει για να είμαι ειλικρινή ή θα έχει μια άμεση νομική δεσμευτική ε, επίδραση που σημαίνει ότι θα πρέπει ίσως να αλλάξουμε τη συνθήκη και κατά την άποψή μου αυτό είναι αδύνατον ή μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια εγώ ακόμα δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, αλλά είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, για το άνοιγμα της οδηγίας για την ε, απόσπαση των εργαζομένων, να σας πω ότι η κυβέρνησή μου είναι αντίθετη σε αυτό και υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο πρώτος είναι ότι εγώ πλέον έχω εξοικειωθεί με την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Μας πήρε χρόνια, δεκαετία νομικής ασάφεια ε, στον τομέα για να καταλήξουμε σε μια λήξη. Και πιστεύω ότι εάν ξεκινήσουμε και ανοίξουμε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων θα έχουμε πάλι δεκάδες χρόνια νομικής ασάφεια και δεν ξέρω αν αυτό θα αποτελέσει λύση. Ε, το δεύτερο είναι ότι φοβάμαι, και εδώ δεν σας μιλάω ως Προεδρεύον του Συμβουλίου, σας μιλώ ως Σουηδός υπουργό Απασχόλησης. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου εάν καταφέρουμε να έχουμε μια αναθεωρημένη οδηγία, θα έχουμε λιγότερη ευελιξία. Και αυτό θα είναι αποτρεπτικό για το σουηδικό μοντέλο. Αυτό αυτό λοιπόν είναι ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Βέβαια το θέμα είναι φλέγον, θα πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί στις συζητήσεις μας με τους κοινωνικούς εταίρους, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και με το Κοινοβούλιο, για να δούμε πώς μπορούμε να μετριώσουμε τις εύλογες ανησυχίες των κοινωνικών εταίρων για το θέμα αυτό. Είμαι Βεβαίω, κύριε Φάλμπρον και κυρία Σρέντερ ότι αυτό δεν σα ικανοποιεί ω απάντηση, αλλά τουλάχιστον εμεί ε, το έχουμε σκεφτεί αυτό το θέμα και προσπαθούμε να βρούμε μία λύση. Κυρία Στρέλα, όπω ξέρετε, όπως είπατε και εσείς, συζητήσαμε πριν από ένα μήνα την οδηγία για την ε, άδεια μητρότητας. Όπως έχουμε συμφωνήσει, θα συνεχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε το θέμα, θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν περισσότερο και φυσικά ως Προεδρία χρειαζόμαστε και στην συνεργασία ε, και με εσά την ίδια αλλά και με όλο το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε λύση. Πιστεύω βέβαια ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, διότι αν δείτε το ίδιο το θέμα, υπάρχουν ε, αποκλίνουσες απόψεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε μία λύση για να προχωρήσουμε. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συνένεση στο Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Έτσι εκλαμβάνω εγώ την κατάσταση, αλλά θα εργαστούμε και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να έχουμε την κατάλληλη ισορροπία για το θέμα. Καλό θα ήταν να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό ε, όσο το δυνατόν συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Κασέφη. Θα θέλατε να κάνετε και εσείς κάποιες ε, διευκρινήσεις ίσως. Απλά θέλω να πω στους συναδέλφους ότι αν θέλετε να μιλήσετε όλοι πρέπει να αυτοπιθαρχηθούμε. Κυρία Κασέφη, θέλετε εσείς σε συντομία να συμπληρώσετε κάτι στις απαντήσεις του Υπουργού ή να ακούσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις και να πάρετε το λόγο στη συνέχεια. Τι προτιμάτε. Να ένα σύντομο σχόλιο θα κάνω για το έτος καταπολέμησης της ε, φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, το 2010 δηλαδή. επεξεργαζόμαστε αυτά τα ζητήματα και η κυρία Πλάμ μας έκανε την ερώτηση αν έχουμε ε, μία στρατηγική για το έτος 2010. Φυσικά έχουμε αρχίσει τις συζητήσεις και η Επιτροπή συνέστησε μια συμβουλευτική επιτροπή προγραμματισμού και συντονισμού των ε, ζητημάτων που θα μας απασχολήσουν το 2010. Θα γίνει διάσκεψη τρογγυλής τραπέζης για το θέμα αυτό και τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν το 2010. Η Σουηδική Προεδρία δε θα κάνει μια ενακτήρια διάσκεψη για αυτό το θέμα και συνεχίζουμε τις συζητήσεις με την Ισπανία για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Αρχίζουμε με το δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ο κύριος Τούσας, παρακαλώ. Και... Η αλλαγή εκπροσώπησης στο επίπεδο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει συνέχεια και έχει μια ευθύνη σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της πολιτικής. Πραγματικά αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε σε ό,τι αφορά τους τομείς που εξετάζουμε σήμερα, μετά αρκετά χρόνια, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας, του 2000 και του 2005 όπως επικαιροποιήθηκε, ενώ σε όλη αυτή τη φάση διαπιστώνεται η διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, από την άλλη διαπιστώνεται δεινά για τους εργαζόμενους. Χθες κύριε Υπουργέ παρουσιάστηκε στην Επιτροπή μας μία μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων μορφών εργασίας στις βιομηχανικές σχέσεις και στην εξέλιξη της εργασιακής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί αποτυπώνεται αυτές, εκεί αποτυπώνονται οι οδυνηρές συνέπειες που έχουν αυτές οι αλλαγές σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους σε θεμελιώδη μισθολογικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Και είναι σωστό να αναφερόμαστε σε ό,τι αφορά στον οικονομικό τομέα. Αλλά εδώ έχουμε μια βαθύτερη, αντιδραστικότερη εξέλιξη σε ένα βασικό σημείο που ο προηγούμενος συνάδελφος ανέφερε επιγραμματικά. Αμφισβητείται πλέον το δικαίωμα των εργατικών συνδικάτων να διαμορφώνουν αιτήματα και το πλαίσιο των διεκδικήσεών τους και το δικαίωμα της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Σε αυτό χρησιμοποιείται το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι γνωστές άλλωστε οι αποφάσεις για την υπόθεση Λαβάλ, Βίκυ Λάινγκς και μια σειρά άλλες στη συνέχεια. Και θέλουμε μια απάντηση σχετικά σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Δεύτερο στοιχείο. Η ανεργία Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο του 2009 εκτινάχθηκε στα 21.794.000. Αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2008 κατά 5.111.000. Η Ισπανία χτυπιέται με ανεργία της τάξης του 18,5%, η Λετωνία με το 17,4%, η Λιθουανία με το 16,7%. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο χειρότερη. Σε ό,τι αφορά τους νέους ιδιαίτερα, που είναι μέχρι 25 ετών, καταγράφεται το, ποσοστό, το γενικό ποσοστό της ανεργίας σε 19,7% με μεγαλύτερο ποσοστό στην Ισπανία 38,4% και στη Λιθουανία με το 30,9%. Ολοκληρώνεται αυτή η φάση και πλέον από το 2010 θα έχουμε τη νέα στρατηγική για την απασχόληση. Είναι προφανές ότι στο Συμβούλιο του Μάρτη θα παρουσιαστεί η σχετική έξεδεση και οι άξονες που θα προετοιμαστούν επί της Σουηδικής Προεδρίας. Ποιες είναι οι γενικές κατευθύνσεις που διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά αυτή την κατεύθυνση. Και να τελειώσω με το τρίτο στοιχείο, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρο, θέλω λίγο την ανοχή σας, για ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Χθε είχαμε την ε, συνάδελφό σας εδώ, την κυρία Μαρία Λάσον, αν λέω σωστά το όνομα, ε, Αγαπητέ συνάδελφοι, αν μπορείτε να ολοκληρώσετε για να έχουμε χρόνο για όλους. Η κοινωνική ασφάλιση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ίδια το επεσημάνε αυτό. Τι έχουμε σε ό,τι αφορά τώρα, ως γενικευμένο παράδειγμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι το εξής. Χαρακτηρίζονται η κοινωνική ασφάλιση ως επαγγελματική ασφάλιση σε κλάδους εργαζομένων, όπως είναι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο στη χώρα μας και αναγκάζονται οι γυναίκες που εργάζονται στο δημόσιο στην Ελλάδα να υποστούν τη χειροτέρεση των όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης αυξάνοντας τα όρια ηλικίας από 5 μέχρι 17 χρόνια. Είναι σωστή πραγματικά μια τέτοια εξέλιξη. Ποιο είναι η ελκυστική πρόταση που πραγματικά προτείνεται σε ό,τι αφορά το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Στίφεν Χιούς και η κυρία Έλντα Φικυρέιδο ακολουθούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτη ερώτηση προς την κυρία Κασέφη αναφέρατε τον κανονισμό 883 του 2004 ε, αναφερθήκατε στη σχετική συμφωνία μπράβο και εμείς ε, χαιρόμαστε για τη συμφωνία αυτή αλλά υπάρχει μια δήλωση με ημερομηνία 20 Ιουλίου του 2009 και όπου λέγεται ότι οι πληροφορίες για τον πίνακα 2 θα πρέπει οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δοθούν ως το δυνατόν πιο γρήγορα ε, δίχως καθυστέρηση ε, ε μετά από αίτηση του σχετικού ε, ιδρύματος και όχι αυτόματα ε, στην τσεχική προεδρία η δήλωση αυτή τελείωνε πριν από το όχι αυτόματα. Ε, τώρα που αναφέρεται το όχι αυτόματα κατά την άποψή μας ανατρέπεται η συμφωνία της τσεχικής προεδρίας θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό δεύτερη ερώτηση έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που θα εφαρμόσετε για το χρόνο εργασίας μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα επίσης για τις αποσπάσεις ε, και, για και μετά την υπόθεση Λαβάλ μπορεί να υπάρχει ε, να έχει επιληθεί το πρόβλημα στη Σουηδία αλλά σε άλλες χώρες του Ηνωμένου Βασίλειου ακόμη κρεμούν ζητήματα και η νομική αβεβαιότητα συνεχίζει να υφίσταται είτε ασχοληθούμε με την οδηγία για τις αποσπάσεις είτε όχι. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία αυτή για να ο, ξεκαθαριστεί ε, το κατά πόσον, ποια είναι τα ελάχιστα όρια και τα ελάχιστα standards τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος, κυρία Φιγκερέιδο. Και μετά ο κύριος ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω τρεις ερωτήσεις που παρότι έχουν ήδη ακουστεί ε, θέλω να τις εμβαθύνω. Πρώτον, στρατηγική της Λισαβόνας. Πολύ σημαντική ανησυχία. Γιατί η αναθεώρηση που έγινε, η ενδιάμεση αναθεώρηση, επιδίνωσε αυτό, αυτή την φιλελεύθερη θεώρηση που επικρατούσε στη στρατηγική της Λισαβόνας. Και σήμερα η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε είναι εντελώς φιλελεύθερη. Γνωρίζετε τις αποφάσεις Ρούφερτ Λαβάλ από το ΔΕΚ που δημιουργούν μέγιστη ανασφάλεια, όχι νομική, αλλά αμφισβητούνται θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και αμφισβητείται το ίδιο το κοινωνικό, ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Οδεύουμε προς ε, μια κατάσταση που σχεδόν μας εξομοιώνησε με χώρες που κοροϊδεύαμε. Λέγαμε ότι η κατάσταση σε αυτές τις χώρες ήταν επιζήμια γιατί δεν προστάτευαν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το ίδιο κάνουμε και εμείς τώρα. Πώς λοιπόν προετοιμάστηκε η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας για να ληφθούν υπόψη αυτά τα προβλήματα κάτι άλλο τώρα. Πώς είναι δυνατόν να συμφιλειωθεί αυτή η ύψιστη προτεραιότητα που είχε αποδοθεί στον ανταγωνισμό με και τις αρχές ε, του συμφώνου σταθερότητας ε, που γίνονται λίγο πιο ευέλικτες, ε, γιατί είπε ο Υπουργός ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη, πώς συμφιλιώνονται αυτό με την ε, οξία επιδίνωση της ε, ανεργίας ε, των χαμηλών μισθών, της αύξησης της φτώχειας, κυρίως όταν πλησιάζουμε το 2010, που είναι το έτος της φτώχειας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Προπάγανδα είναι. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε την κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε τους εκπροσώπους της ε, Σουηδικής Προεδρίας στις παρεμβάσεις σας. Μου δώσατε την εντύπωση ότι είστε ε, πολύ αισιόδοξοι. Είπατε ότι είναι προσωρινή η κρίση και ότι δεν ε, θα διαρκήσει εσάι. Όμως πολλοί αναλυτές ε, πρεσβεύουν ότι θα είναι μόνιμη η κρίση, πάγια. Ε, βλέπουμε την ανάκαμψη όμως μέσα σε αυτή την κατάσταση των ΗΠΑ και ε, φοβάμαι ότι θα πληγεί πολύ πιο ισχυρά η Ευρώπη. Έχετε κάποιο εφεδρικό σχέδιο, το περίφημο Plan B, τι θα γίνει αν δεν τα καταφέρουμε, τι θα γίνει με την εργατική νομοθεσία. Χρειαζόμαστε τέτοιο εφεδρικό σχέδιο. Thank you. Uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τούσα, μόλις πήρα ένα αντίγραφο των εκθέσεων και έχω διάβασμα απόψε. Οι εμπορικές, οι βιομηχανικές σχέσεις. Πιστεύω ότι λόγω της κρίσης είναι θεμελιώδη σημασία όχι μόνο να έχουμε εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, αλλά και ενεργό συμμετοχή τους σε κάθε πτυχή. Διότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε μια κάποια αξιοπιστία και πώς να σας το πω, κάποια κοινά στοιχεία στη συνεργασία μας και στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανά την Ευρώπη αλλά και ανά την ιστορία. ο αποκλεισμός ε, των κοινωνικών εταίρων ε, και κατά τη διαχείριση της κρίσης ενεργά αλλά και στις ε, βιομηχανικών σχέσεων, τελικά μας οδήγησε σε σκοτεινά μονοπάτια. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα και από μια περιοχή η οποία υπερηφανεύεται ότι έχει καλό κλίμα εργασίας και συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους. Και ως αποτέλεσμα, αν ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες του κόσμου, οδήγησε σε πολλά πράγματα και σε λιγότερες ε, συγκρούσεις. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδους σημασία ε, για ένα καλό εργασιακό κλίμα και φυσικά για να μπορέσουμε να επανακάμψουμε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις βραχυπρόθεσμες κρίσεις, αλλά και μακροπρόθεσμα να προσαρμαστούμε στις υφιστάμενες συνθήκες, αν θέλετε. Εγώ προέρχομαι από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση βέβαια, αλλά αυτό δεν έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι πρέπει να συνάγουμε συμπεράσματα από το γεγονός Ε, και το βασικό συμπέρασμα είναι ότι χρειάζεται να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Την έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντικό να τη διαβάσω. Ε, εν μέσω κρίση συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα και φυσικά πρέπει να επανέλθουμε. Θα επανέλθω και στην ε, υπόθεση Λαβάλ σε λίγο ε, την αύξηση της ανεργίας. Ναι, είχαμε 2% αύξηση της ανεργίας ε, από την προηγούμενη χρονιά πέρσι. Αυτά είναι τα στατιστικά στοιχεία του Ιουλίου. Αυτό είναι φυσικά πολύ σημαντικό και θα ε, επιβαρύνει όλα τα ε, κοινωνικά συστήματα ασφάλισης στην Ευρώπη. Ο αποκλεισμός ε, από την αγορά εργασίας ήταν υψηλός ούτως ή άλλως κατά την άποψή μου πριν ενταχθούμε στην κρίση. Και η ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων είναι το βασικό πρόβλημα. Έχουμε έχουμε όμως και άλλα περιστατικά ε, κοινωνικού αποπλισμού. Προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε, για παράδειγμα, την ε, οικονομική κρίση τη δεκαετία του 90 και οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την κάλυψη των ε, συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και είπαν ότι αυτή ήταν η αιτία που δεν μπόρεσαν να επανακάμψουν στην αγορά εργασίας. Και φυσικά αυτό επιβάρυνε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Φυσικά και θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε στενά και να βρούμε μία λύση. Και οι δημόσιε χρηματοδοτήσει ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και εδώ έγινε και το θέμα της ισορροπίας. Αν δεν έχετε καλά δημόσια οικονομικά, δεν θα μπορείτε να πληρώσετε για τα αποτελέσματα της κρίσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και όταν αρχίσει να περνάει η κρίση. Για να είμαι ειλικρινής, είναι σαν τους Κινέζους ε, καλλιτέχνες ε, του τσίρκου που έχουν 5-6 ε, μαστίγια ή ξυλαράκια ταυτόχρονα και προσπαθούν να τα ε, χρησιμοποιήσουν όλα ταυτόχρονα, σαν τους ζογκλέρ. Έτσι είναι η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Και εκεί φυσικά ε, είναι που πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε και να βρούμε λύσεις. Και αυτό ήταν από τα βασικά θέματα του άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου τον Ιούλιο, στις αρχές Ιουλίου. Ένα συνδυασμό λοιπόν δράση, παιδεία και μείωση των κατοφλίων ε, για τον νέων για να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας είναι από τα βασικά ε, θέματα που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και να συνεργαστούμε. Κύριε Χιούς, η, ε, οδηγία για το χρόνο εργασίας. Στις αρχές Ιουλίου στο Άτυπο Συμβούλιο κάναμε και μια σύντομη συζήτηση, μόλις είχαν σταματήσει και οι διαπραγματεύσεις και προσπαθούσαμε να δούμε πού είμαστε. Δεν είμαι τόσο αισιόδοκτο, ε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα δεν φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσει στο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει το δύσκολο καθήκον να προσπαθεί να βρει ε, μια λύση, ένα δρόμο να προχωρήσει και ε, είμαι Απεσιόδοξο για να σα πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Η θέση στο Συμβούλιο δεν έχει αλλάξει. Τα, πρόβλημα τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται σε πολλές χώρε μέλη και κατά την άποψή μου θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Οι ανησυχίε που ακούσαμε ε, υπάρχει και η επιλογή του opt-out ε, και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αλλά δεν είναι εύκολο να βρούμε μια ισορροπία που θα ικανοποιήσει και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε, αποκινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προσπαθήσουμε να βρούμε αυτή την ισορροπία ε, και για να είμαι ειλικρινή πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ επικοδομητικοί και να έχουμε συνεχώ επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφύγουμε περαιτέρω κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο επόμενο στάδιο. Τώρα, για την υπόθεση Λαβάλ. Όταν εγώ παρουσίασα Το αποτέλεσμα της έρευνας ε, στην αρχή του ε, Συμβουλίου τον περασμένο Δεκέμβριο δεν υπήρχε ούτε ένα κράτος μέλος στο Συμβούλιο που ήταν ε, διατεθειμένο να ξανανοίξει την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Ταυτόχρονα κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα και κατανοούμε και ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανοιχτόμυαλοι σε συζητήσεις, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό. Όπως σας είπα, ε, εγώ ξεκίνησα στην υπόθεση Λαβάλ από το γεγονός ότι μας δυσαρέστησε ιδιαίτερα το αποτέλεσμα της, ε, του δικαστηρίου και μετά είχαμε και τη υπόθεση του Λουξεμβούργου. Ε, όλα αυτά ήταν δυσάρεστα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτόμυαλοι στη συζητήση με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν υπάρχουν άλλε δίωδοι. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά ξεκίνησε μια διαδικασία με περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη διαφάνεια και θεωρώ ότι αυτά είναι καλά αρχικά μέτρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφός σας ε, ε, είναι δυσαρεστημένος, ε, θα το ελέγξω. Κυρία Φιγκερέιδο, συγγνώμη δεν μπορούσα να προφέρω το όνομά σας. Η στρατηγική της Λισαβόνας είναι κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολύ στενά με την ε, ε, μελλοντική Ισπανική Προεδρία και ελπίζουμε να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε συμπεράσματα το Δεκέμβριο, τα οποία θα αποτελέσουν και τον ακρογωνίο λίθο για τη συνέχεια τη δουλειά τη Ισπανίας. Όπω σα είπα, εγώ εκπροσωπώ μια κεντροδεξιά κυβέρνηση στη βόρεια κυβέρνηση και ο συνάδελφο μου από την Ισπανία εκπροσωπεί μια σοσιαλιστική κυβέρνηση από την Νότια Ευρώπη και συνεργαζόμαστε πολύ καλά και αυτό είναι πολύ καλό μήνυμα. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε και στην ε, παρούσα και στη μελλοντική στρατηγική της Λισαβόνας είναι πώς μπορούμε να τη συγκεράσουμε και να έχουμε ένταξη, εκπαίδευση, να επανεντάξουμε τους ανθρώπους στην αγορά εργασία, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα συστήματα που έχουμε, πολλά από τα οποία είναι εκτός του δικού μου του πεδίου, για να μπορέσουμε να ε, ξαναστήσουμε την Ευρώπη στα πόδια της. Και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας ε, για το θέμα αυτό. Κυρία Γιακονσάρη, η συνάδελφος από τη Φιλανδία. Ένα εφεδρικό σχέδιο είπατε. Εγώ έχω μάθει ότι πάντα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ένα, αλλά και ένα δεύτερο και ένα τρίτο εφεδρικό σχέδιο. Διότι η ιστορία ποτέ δεν επαναλαμβάνεται και ποτέ δεν έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που νομίζαμε ότι θα έχουμε στην αρχή. Τα πράγματα αλλάζουν και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Ποιος θα φανταζόταν, ας πούμε, πέρσι ότι θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε τώρα. Απ' την άλλη, πριν από έξι μήνες ε, όλοι μιλούσαν για μια οικονομική διάλυση και υπήρχαν προγνώσεις ε, για πραγματικό κράχ. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε λίγο διαφορετικές ε, περιστάσεις. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα. Θα πρέπει να ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά του συναδέλφου και να προσπαθήσουμε να βρούμε την κατάλληλη λύση από αυτά που λένε και να είμαστε και ανοιχτόμυαλοι και να αλλάζουμε αυτά που πρέπει να αλλάζουν. Ε, μιλάω σαν Ινδός γκουρού εδώ, ε, δεν προσπαθώ να κάνω το, τον έξυπνο εδώ, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και να τα παίρνουμε λίγο πώς έρχονται και να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι με αυτά που έχουμε. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, το πρόγραμμα ανάκτησης, ε, ανασύστασης, ε, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε επίσης να έχουμε ένα ασφαλές ε, οικονομικό σύστημα να την Ευρώπη για να μπορέσουν να προχωρούν και οι επιχειρήσει μα και ταυτόχρονα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε την ε, ανεργία λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορούμε να σώσουμε όλες τις θέσεις εργασίας, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε το εργατικό δυναμικό μας. Μπορούμε να έχουμε περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη ε, ενεργό συμμετοχή. Το ξέρω ότι δεν είναι η τέλεια απάντηση, αλλά δουλεύουμε με αυτά που έχουμε. Ευχαριστώ. Thank uh, <clears throat> uh, Θα ήθελα να αρχίσω με την, τις παρατηρήσεις του κυρίου Τούσα. Επιβεβαιώνω αυτά που είπε φυσικά χτες η Μαρία Λάρσον Ότι δηλαδή είναι θέματα εθνικής αρμοδιότητας αυτά που συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση και τις παροχές. Φυσικά δεν έχουμε καμία πρόθεση να αλλάξουμε την κατάσταση. Για την ε, μετά την ε, Λισαβόνα διαδικασία, Έχει γίνει συζήτηση για την ενεργοκοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι παραδοσιακά η πολιτική απασχόληση βασίζεται σε ενεργά μέτρα. Δυστυχώ, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική ασφάλιση, μάλλον παθητική στάση τηρούμε. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Και δεν μιλάμε για αύξηση της οικονομικής ασφάλειας των ε, ανθρώπων ε, ή να συνταξιοδοτούνται οι άνθρωποι νωρίτερα. Το αντίθετο, ε, λόγω της δημογραφικής κατάστασης στην Ευρώπη θεωρούμε ότι πρέπει να εισέρχονται νωρίτερα στην αγορά εργασίας οι άνθρωποι, να εργάζονται περισσότερες ώρες και να απέρχονται αργότερα. Ε, και θέλουμε για να το πετύχουμε αυτό μια, να, να πετύχουμε μια υγιέστερη ζωή στην αγορά εργασίας και μια καλύτερη κοινωνική ασφάλιση. Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για αυτά που μας είπε ο κύριος Χιούς. Μάλιστα, υπό τσεχικής προεδρίας υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δεν προετοιμάζουμε τώρα επίσημη απόφαση. Ξέρετε, κύριε Χιούς, είναι εξαιρετικά περίπλοκο και τεχνικό το ζήτημα. Ελέγχουμε να δούμε αν υπάρχουν λάθη στην εφαρμογή της νομικής ε, πράξης και θα επανέλθουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ ε, επειδή δεν αυτοπιθαρχήθηκε κανένας, φτάνω στο δύσκολο σημείο τώρα να μειώσω το χρόνο αγόρευσης σε 1,5 λεπτό. Ζήτω συγγνώμη. Γιατί αλλιώς δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις των Υπουργών. Η κυρία Ελίζαμπεθ Λίν, λοιπόν, 1,5 λεπτό παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που είπατε ότι δεν ε, πρέπει να αποκλείεται κανείς από την αγορά εργασίας πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο να μπει να συμμετάσχει στην αγορά εργασίας ε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό πρέπει να σκεφτούμε αν και εφόσον υπάρχει ορισμός της αναπηρίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να δουλέψουν πρώτη ερώτηση αυτή ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω αναπηρίας, λόγω θρησκείας, λόγω ε, ηλικίας αποκλείονται την σημερινή μέρα από την ε, αγορά εργασίας. Είναι εμείς θα θέλαμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Σας παρακαλώ λοιπόν να μου, μου κάνετε τα σχόλιά σας. Η κυρία Μαρίτα Ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα, γιατί δεν είμαι τακτικό μέλος ε, της Επιτροπής. Εγώ απλώς αντικαθιστώ ένα τακτικό μέλος της Επιτροπής. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Λιτορίν και την κυρία Κασέφη Γιατί βλέπω ότι άφησε και μουσάκι ο κύριο ε, Λιτορίν. Ε, ε, και περίμενα να, τον περίμενα σαν να η Βασίλη να μας φέρει και κάνα δωράκι, αλλά στεναχωρήθηκα τελικά, δεν μας έφερε τίποτα. Έχουμε την απόφαση Λαβάλ, την απόφαση Βίκινγκ, τη, στο Λουξεμβούργο. Τελικά έχουμε μια οδηγία de όχι de minimis. και τελικά παρεμποδίζει την ίση μεταχείριση των μισθωτών στην Ευρώπη. Η κυρία Κασέφη μας μίλησε για ισότιμη μεταχείριση μέσα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μα αυτό δεν ισχύει στην αγορά εργασία. Ε, λόγω, εξαιτία αυτή τη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Όταν έρχεται κάποιο από μία άλλη χώρα και πάει σε ένα άλλο κράτο μέλο να εργαστεί, δεν ισχύουν οι ίδιες συνθήκες, δεν ισχύουν τα ίδια δικαιώματα. Ε, αυτά, ε, και παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονικά ε, έπρεπε να τηρούμε απαρέγκλητα αυτούς τους όρους τώρα λόγω της κρίσης. Στην ε, Σουηδία τα συνδικάτα δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις. Πίεση δέχεται και η αγορά εργασίας και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η, αν πάρα πολύ γρήγορα η ανεργία, παρακαλώ ε, ε, θα ήθελα να κλείσετε την παρέμβασή σας. Μα θέλω να κάνω μια ερώτηση, μα δεν προλαβαίνετε, έχετε εξοδέψει το χρόνο αγορασή σας. Ένα μισή λεπτό είπαμε, συγγνώμη. Τελείωσε ο χρόνος σας, καταλαβαίνετε. Δηλαδή μπορώ να θέσω την ερώτησή μου. Ο κύριο ευχαριστώ. Ακούσαμε ευσεβεί πόθου, ωραίου στόχου, ωραίε φιλοδοξίε. Όλοι θέλουν απασχόληση, όλοι θέλουν να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, όλοι θέλουν βιώσιμε αγορέ εργασία και μεγάλη απασχόληση. Μα πώ θα το κάνετε αυτό. Και άρχισα να σημειώνω. Ο κύριο Λιτόριν θα αρχίσει τι συζητήσει. Η κυρία Κασέφη άρχισε ήδη τι συζητήσει και θα υποστηρίξει τη συνέχεια των συζητήσεων. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε, θα κάνουμε σεμινάρια. Πάω από με έχετε Πολύ ωραία πολιτική έχουμε. Πολύ ενεργό η πολιτική σα. Η ανενεργή πολιτική πώ θα ήταν δηλαδή. Άμα μου τα είχατε πει αυτά πριν από 5-10 χρόνια, τα ίδια θα ήταν και άμα ξανάρθουμε τώρα σε 5-10 χρόνια πάλι τα ίδια θα μας λέτε επί της ουσίας. Ε, ποια ουσία δεν υπάρχει ουσία. Μιλάτε για το συντονισμό για τους υπηκόους τρίτων χωρών μάλιστα μάλιστα. Τίποτα ουσιαστικό δεν μας είπατε. Τι θα πετύχετε μπορείτε να μας πείτε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Πρέπει να μειώσουμε τα αντικίνητρα για τους εργοδότες, να μειώσουμε τους φόρους ε, για την ε, σε εργασιακούς φόρους ε, και αυτό μόνο θα αυξήσει τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Ε, ουσιαστικά οδόφραγμα είναι το, η πολιτική σας. Ε, δεν ε, βοηθάει την εκπλήρωση των στόχων που μας παρουσιάσατε. Πώς θα γίνει πιο ευέλικτη η, ομάδα, ε, η αγορά εργασίας. Πώς, ποια θα είναι τα κίνητρα για τους εργοδότες για να φέρουν περισσότερους μέσα στην αγορά εργασίας. Τίποτα σχετικό δεν μας είπατε. Σας ευχαριστούμε που σεβαστήκατε το χρόνο αγόρευση. Ο κύριος Σέρκας, τελευταίος ομιλητής αυτό το γύρο. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε και για τη διαλεκτική σας ικανότητα. Πολύ τηλεγραφικά δύο-τρία πράγματα. Για την κοινωνική ρήτρα να σας πω ότι αυτή θα ήταν μια έξοχη ε, δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε μια ε, συνθήκη της Λισαβόνας που θα ανταποκρίνεται σε πολλά από τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας, δικαιώματα για τους εργαζομένους. Επομένως αυτή είναι μια καλή οδός. Για την υπόθεση Λαβάλ δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν είναι δύο-τρεις υποθέσεις, δεν είναι μερικές εκατοντάδες, είναι εκατομμύρια των εργαζομένων αυτοί που ανησυχούν, διότι χάθηκαν οι αρχικοί στόχοι τη οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση, υπάρχουν κάποια ελάχιστα τα οποία μετατράπηκαν σε μέγιστα. Υπάρχει λοιπόν μια σοβαρή νομική ανασφάλεια, δεν είναι ε, το άνοιγμα τη οδηγία ε, αυτό που δημιουργεί νομική ανασφάλεια, αλλά είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τη συμμετρία μεταξύ των αρχικών στόχων και το αποτέλεσμα τη απόφαση του δικαστηρίου. Αυτό που έκανε η απόφαση του δικαστηρίων ήταν να δημιουργήσει μια τεράστια ε, νομική και πολιτική ασάφεια και θα ήθελα να ξέρω ε, τι ακριβώς μπορεί να κάνει το σουηδικό κοινωνικό μοντέλο για να αλλάξει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, την ίση εργασία για όλους. Και κυρία Κασέφη, το 2010 έχουμε όντως ε, το έτος κατά την ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ελπίζω στην Ισπανική Προεδρία να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μην κάνουμε αυτό που είπε και ο προλαλής σας, να μιλάμε χωρίς να έχουμε πράξεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λίνα, θα ε, μιλήσω για τον ορισμό της αναπηρίας σε λίγο, αλλά ε, την κυρία Ουλτσκοφ, η οποία ήταν τέλος γενική γραμματέας του διαφορετικού κόμματος βεβαίως, τα, την κυρία Ουλσκόφ λοιπόν τα θέματα τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Ε, άλλο βέβαια το εθνικό πλαίσιο και άλλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο με την με το παλιό νομικό πλαίσιο που είχαμε ε, μπορούσαμε να αποκλείσουμε και να μην λάβουμε υπόψη μας ξένη αλλοδαπή συλλογική σύμβαση. Τώρα, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, δεν λέγεται ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, να αποκλείσουμε, αλλά τα πράγματα είναι πιο φλού, αν θέλετε. Ε, άρα τα, η υπόθεση είναι περίπλοκη και βεβαίως θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις, γιατί ε, ε, και που δεν είναι λόγο θα σταματήσει η συζήτηση για το θέμα αυτό γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πράγματα ακόμη κρεμούν και η νομική αβεβαιότητα είναι μεγάλη. Αλλά υπάρχουν και υπάρχουν και βεβαίω, αν δεν υπήρχε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα είχαμε τον χρόνο να κάνουμε άλλα πράγματα. Ε, θα, θα δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία, πιο μακροπρόθεσμου στόχου κτλ. Κύριε Χέλμερ. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σα και το θυμό σα Σε ευρωπαϊκό επίπεδο προφανώς δεν ε, έχουμε τόσα πολλά εργαλεία ο, στα χέρια μας. Ε, εδώ υπάρχουν και εθνικές αρμοδιότητες. Διαφωνώ ωστόσο μαζί σας με αυτό που είπατε ότι εδώ απλώς λέμε ωραία λόγια. Όχι. Στα σε κάποια κράτη-μέλη εφαρμόζονται μέτρα πολιτικές ε, που ε, μειώνουν αν θέλετε τον κοινωνικό αποκλεισμό και στη δική σας τη χώρα και σε τούτη και στη δική μου τη χώρα έγιναν πράγματα και μεγάλος αριθμός αποκλεισμένων κοινωνικά ατόμων επανήλθαν στην αγορά εργασίας. Επίσης έγιναν αλλαγές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, αυξήθηκαν επιδόματα, ε, ορίστηκαν διαφορετικά κατόφλια όπου κάποιοι ε, ε, βγήκαν ας πούμε από τη σύνταξη αναπηρίας που έπαιρναν και μπήκαν σε ένα άλλο σύστημα πιο αποδοτικό για αυτούς. Ε, ού μόνον σε ένα σύστημα συνταξιοδότηση πιο αποδοτικό για αυτού, αλλά μερικοί και στην αγορά εργασία. Υπάρχουν προκλήσει πάντως και τι προκλήσει αυτές θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε και ε, προφανώ πρέπει να μάθουμε η από του δε διαφορετικά η Ευρώπη δεν λειτουργεί. Τέλο κυρία Σέρκα, όντω πιστεύω ότι στην μετάφραση μετά Λισαβόνα εποχή θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να δούμε πιο συγκεκριμένα πώς μπορούμε να επαναφέρουμε κόσμο στην αγορά εργασίας και δει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό. Ε, η έρευνα και η ανάπτυξη είναι ένα που πρέπει να τον δούμε ε, να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Δεν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά βεβαίως. Ε, και εγώ πολλές φορές εκνευρίζομαι και θυμά, θυμώνω. Γιατί βεβαίως συνεχώς μας ρωτούν και τι κάνατε, πού είναι ο Άγιος Βασίλης, τι μας έφερε δωράκι ο Άγιος Βασίλης και δεν έχω πολλά πράγματα να απαντήσω. Λάβετε όμως υπόψη σας ότι η στόχη αυτή είναι δύσκολο να επιτευθούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν και διαφορετικά μέτρα και εργαλεία ε, στα διαφορετικά κράτη-μέλη. Ωστόσο έχουμε κάποια στοιχεία από την πείρα μας, ο καθένας από τη χώρα του, που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Madam Chair. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει και η κυρία Κασέφη. δεν θα συμπληρώσω τίποτα σε αυτά που είπε ο κύριος Λιτόριν ε, για την παραφορά τόμων αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας κτλ. Εγώ θα αναφερθώ στο θέμα της αναπηρίας, disability. Ε, υπάρχει θέση του Συμβουλίου, μια πρόταση, εν πάση δεν υπάρχει συχνόν πρόταση στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό και η Προεδρία δεν έχει προγραμματίσει να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Sorry, it was your views on a new directive in access to goods and services that the Parliament voted for. Which... Μα στην οδηγία για τα εμπορεύματα και τις υπηρεσίες ε, που προτείνατε εσείς εμπλέκεται και η έννοια της αναπηρίας. Θα ήθελα λοιπόν να δω τι κάνετε με αυτή την οδηγία γιατί εκεί μπορεί να μπει το θέμα του ορισμού της αναπηρίας. Yes, I'm sorry. Uh, ναι, συγγνώμη. Αυτή η οδηγία δεν είναι της αρμοδιότητάς μας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να κρατήσουμε σημειώσεις και να επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να σας υποσχεθώ. Θα μιλήσουμε όμως για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε να μας το διαβάσετε για να ενημερώσουμε και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής. Ελιζαμπέτ ε, Μογά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, μάθω ποια είναι η θέση της Σουηδικής Προεδρίας ε, για την συνέχιση που θα δοθεί στις εργασίες για την προσωρινή εργασία. Είναι δύσκολη κατάσταση και η ευελιξία που αναμένουν διάφορες επιχειρήσεις από τους εργαζομένους καθιστούν επισφαλέστερη την κατάσταση. Πέρσι, στο τέλος του χρόνου, ελήφθη μια απόφαση για την προσωρινή εργασία και Έχετε εσείς αποτελέσματα μελετών για να δούμε σε ποια ε, κατάσταση έχουν περιέλθει όσοι εργάζονταν ε, με αυτό το καθεστώς. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τούρινεν, ευχαριστώ τους υπουργούς ε, για την παρουσίασή τους. Πολλοί ε, ξαφνιάζονται με την απάθεια που επικρατεί παρά την αύξηση της ανεργίας και την επιδείνωση της κοινωνικής κατάστασης πώς γίνεται και έχουν εκλείψει όλες οι κοινωνικές ε, πρωτοβουλίε γιατί δεν έχουμε στόχους για να απαλύνουμε τη... τα βάσανα των ανθρώπων. Άκουσα αυτά που μας είπατε. Μιλήσατε για περαιτέρω κατάρτιση, μιλήσατε για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, Μιλάτε για τις εθνικές λύσεις που έχουν υιοθετηθεί στη Σουηδία. Μα δεν μιλάμε τώρα για τα δικά σας εθνικά προβλήματα, μιλάμε για τα ευρωπαϊκά προβλήματα και εφόσον προεδρεύετε στο Συμβούλιο εκ μέρου όλων, Καλό θα ήταν και να ξαναδείτε την οδηγία για την απόσπαση και δεν νομίζω να καταστραφεί έτσι το ισοειδικό μοντέλο. Το αντίθετο μπορεί και να σωθεί. Ε, υπάρχει μεγάλη ανεργία στους νέους. Το βλέπουμε σε όλες τις στατιστικές. Τι θα κάνετε για τους νέους για να ε, μην χαθεί μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Νάρκιν και, και η κυρία Ντανούτα Ζεσλόβγικα. Η κυρία Ζαζλόβιεκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ Λιτουρίν, μιλάμε για τη γύρανση του πληθυσμού και την ε, επέκταση του χρόνου εργασίας. Ε, του ε, όριου συνταξιοδότησης, μάλλον του ηλικιακού όριου συνταξιοδότησης. Ε, εσείς στη Σουηδία είχετε πολύ καλά αποτελέσματα στην αγορά εργασίας και στην εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης. Τώρα, δεδομένης της κρίσης, έχετε κάποιες ιδέες για να βελτιώσετε τα εργαλεία που υπάρχουν για να βελτιωθεί η κατάσταση για τους νέους. Ευχαριστούμε κυρία Εσάγια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργή, μιλήσατε για την ένταξη όλων στην αγορά εργασίας, ακόμη και των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, με αναπηρίες. Ενίοτε, είναι δύσκολο να περάσει κανείς από το πλέγμα της κοινωνικής ασφάλισης, των παροχών, του μισθολογίου, της δομηματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα τι μπορείτε να κάνετε εσείς για να βελτιώσετε την κατάσταση των ατόμων ε, με αναπηρίες ε, μέσα στις ε, επιχειρήσεις. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ισχυρή νομοθεσία, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Παραδείγματο χάρη διατήρηση παροχών, ενώ εισέρχεται αυτό το άτομο μέσα στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν ε, ε, για την πρώτη σας ερώτηση θα συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Κυρίως για την ε, προσερινή εργασία, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, να τους ε, μεταχειριζόμαστε με τον ίδιο τρόπο όπως τους υπολείπους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια λύση. Η ερώτηση της κυρίας Τουρούνεν για το τι ακριβώς κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να απαντήσω ε, με δύο πτυχές. Το ένα είναι το πρόγραμμα ανασύστασης ε, και το άλλο είναι κάτι το οποίο είναι εκτός της αρμοδιότητές μου. Έχει να κάνει με το ΕΚΟΦΗΝ και τους υπουργούς που προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τα δημόσια οικονομικά μας, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ε, υπάρχει κάποια ελπίδα για την οικονομία. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι είναι πολύ λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ξαναέχουμε ε, την εμπιστοσύνη των πελατών στην οικονομία. Και εμείς εγώ προέρχομαι από μια μικρή ανοιχτή οικονομία με το, πάνω από το 50% του ΑΕΠ στο εμπόριο και στις εξαγωγές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εξαρτώμεθα άμεθα με αυτά που, από αυτά που συμβαίνουν έξω από τη χώρα μας Και αυτό νομίζω ότι είναι και ο κανόνας για τι περισσότερε χώρε Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα χαπάκι που μπορούμε να πάρουμε και να τα λύσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στην ε, Ευρώπη υπάρχουν ε, αυτόματοι σταθεροποιητές που τείνουν να εξαφανίσουν κάποιες από τις ε, συνέπειες για τα άτομα μεμονωμένα, παραδείγματος χάρη εντός του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και υπάρχουν και άλλες χώρες ανά τον κόσμο που δημιουργούν dumping στην κατάσταση και θα πρέπει να προχωρήσουμε και πιο ενεργά σε θέματα όπως είναι η παιδεία, και η ενεργοποίηση των ανέργων μας. Για τους νέους, η κυρία Ρουτούρουνεν ρώτησε τι κάνουμε για τους νέους, συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για κοινή ευρωπαϊκή δράση στις συνθήκες μας και στο πλαίσιο βάσει το οποίο εργαζόμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και θα κάνουμε είναι να δούμε τις δράσεις κάθε χώρας και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Μπορεί να είναι απογοητευτικό αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Κατά την άποψή μου, υπάρχουν καλά και κακά νέα για το θέμα αυτό, για τους νέους δηλαδή και... Ε, αυτό που ρώτησε η συνάδελφος από τη, Φιλανδ... Ε, από την ε, Πολωνία η οποία αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Τα καλά νέα είναι ότι η ανεργία των νέων τίνει να είναι μικρότερο χρονικού διαστήματος από την ανεργία των ε, μεγαλύτερων. Αυτό είναι καλό διότι ε, μπορούμε μέσω της εκπαίδευσης ε, και της ενεργοποίησης να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να μην έχουμε μακροπρόθεσμη ενεργία και μακροπρόθεσμο αποκλεισμό. Αυτά είναι καλά νέα φρονώ ότι σε τέτοιους χαλεπούς κυρίους που έχουμε οικονομική κρίση, οι επενδύσεις, οι περαιτέρω επενδύσεις ε, στην παιδεία, στην κατάρτιση και σε τέτοιες μορφής πράγματα είναι υψή τη σημασίας και νομίζω ότι είναι και η καλύτερη επένδυση. Όταν ε, ε, θα βγούμε από την κρίση θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα προετοιμασμένους ανθρώπους που θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την αύξηση της παραγωγής ε, που προσβλέπουμε για το μέλλον. Η κυρία Εσάια ρώτησε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει τα πράγματα. Αναφέρθηκα σε αυτά τα πράγματα, σας είπα και πριν, δεν υπάρχει ένα γρήγορο χάπι. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μέσα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί να ακούγεται απογοητευτικό για πολλούς από εμά, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, και εδώ νομίζω Κύριε Χέλμερ, ε, πριν ε, εκφράσατε την απογοήτευσή σας για το τι μπορούμε να κάνουμε, νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να ανταλλάξουμε τις καλές και τις κακές μας εμπειρίες. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις ε, στις οποίες πήγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα εργαστήριο στο οποίο κάναμε το αντίθετο. Συζητήσαμε τα χειρότερα παραδείγματα και τα χειρότερες εμπειρίες που είχαμε. Και κάποιοι συνάδελφοι από άλλες χώρες ήταν πολύ ανοιχτοί για τα σφάλματα που διαπράξανε. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να μάθουμε ένα από τον άλλον από τα ασφάλματα που έχουμε διαπράξει και να μην τα ξανακάνουμε. Το δει Μαρτίν, άλλωστε. Εργαζόμαστε πολύ στενά σε θέματα εργασίας και θα πρέπει να, με κάθε κόστος να αποφύγουμε την μεταφορά των μακροπρόθεσμα ανέργων σε συντάξεις αναπηρίας, ε, και να μην χρησιμοποιούμε το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης ω ένα μόνιμο πάρκινγκ, χώρο παρκαρίσματος που μπορούμε να του αφήνουμε εκεί και να του πληρώνουμε SAE. Ε, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστώ. Euh, εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ε, η συζήτηση που έγινε ήταν αρκετά πυκνή. Ε, συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα. Μας δώσατε τις απαντήσεις σας. Ε, ε, Έχετε αναλάβει δέσμευση να απαντήσετε στο ερώτημα της κυρίας Λίν για τη μη διάκριση, για τις μη διακρίσεις, για την ίση μεταχείριση. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, έφτασε η ώρα να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Και έτσι προχωρούμε στο σημείο 10 της σημερινής διάταξης που είναι ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό 2010 σας προτείνω Μάλλον να πω ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ήταν να το συζητήσουμε χτες, το, δεν το συζητήσαμε, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Ας κάνουμε πρώτα την ψηφοφορία όμως, ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ε, λοιπόν, ξεκινούμε για το σχέδιο προϋπολογισμού. Έχουμε τον, την τροπολογία 6300. Ποιος είναι υπέρ. Περσόν. Ουδείς. 1300. Υπέρ εκ του 6300. Ε, υπέρ κατά εγκρίνεται. Λοιπόν, 601 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6348 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-16 του Στίβεν Χιούζ απεσύρθη πάμε στο 63-31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-04 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-32 υπέρ κατά αποχές 6306 63-06 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-30 της κυρίας Φιγκερέιδο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63-35 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 07 αυτή καταπίπτει 6308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προχωρούμε στην 6338 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροποποίησης παρατήρησης υπέρ, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 39 του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και άλλη ε, για την παρατήρηση τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή η τροποποίηση 63 17 απεσύρθη της κυρίας Φιγκερέιρο 63-28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-40 καταπίπτει και πάμε στην 63-18 του κυρίου Στίβεν Χιούς α όχι απεσύρθη προχωρούμε λοιπόν 63-29 Φιγκερέιρο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 6309 και 6306 των εισηγητών και Βιντσέντσο Ιεβίνα υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται προχωρούμε τώρα στο 6319 του κυρίου Στίβεν Χιούς απεσύρθη 6341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-20 Στίβεν Hughes υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63-10 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-21 απεσύρθη 63-50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-22 Στίβεν Hughes υπέρ Vous l'avez retiré Alors, il, est retiré. Απεσύρθη. Συγγνώμη. 63-12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63-42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63-43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε τροποποίηση της παρατήρησης ποιος είναι υπέρ. Πρότασή σας κατά αποχές εγκρίνεται 63-11 της υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρα δεν ψηφίζουμε για το σχόλιο 63-44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, προσθήκη προτείνεται στο σχόλιο Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-15 υπέρ η 63-15 και η 63-27 είναι ολόιδιες λοιπόν ψηφίζουμε ποιο ε, ποιος υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 63-25 Στίβεν Χιούς και κυρία Γκόντς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στα 325 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σαφώς με συγχωρείτε 6302 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε για το, το 6302 να γίνει έλεγχος ηλεκτρονικός παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Tout le monde a Έχετε όλες τις κάρτες σας. Mais, que ça marche Mais normalement, ça marche. Réessayez. Mettez votre carte dans le bon sens. Mettez votre... Γυρίστε την κάρτα σας. Βάλτε τη σωστά. Il faut mettre sa carte dans ce sens-là. Hein? La puce vers vous. Tout le monde a pu voter Ωραία, ψηφίσατε όλοι. Μήπως υπάρχει κάποιος που δεν έχει την κάρτα του μαζί.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 Λοιπόν, κύριε Κάστλερ, ψηφίζετε κατά. Να τα σημειώσουμε αφού δεν μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Και ποιος άλλος. Κυρία Βίρ, υπέρ ψηφίζετε. Ωραία. Très Λοιπόν, ωραία, πέρα τις ψηφοφορίες. Donc, il y 39... Εψήφισαν 39, 24 υπέρ, 17 κατά, αποχές 0, Εγκρίνεται λοιπόν η 6302. Καλά κάναμε και κάναμε τον έλεγχο. Προχωρούμε στην 6303 η οποία απεσύρθη. 6313 υπέρ. Ποιος είναι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 6314 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6347 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63-46 του εισηγητή πάλι κατά αποχές εγκρίνεται κυρία εκτός μικροφώνου Which one? Um, 6302 ε, η 6302 έχει μια παρατήρηση, ένα σχόλιο το οποίο πρέπει να δούμε. Ωραία, λέει η πρόεδρος, ναι, ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να ψηφίσουμε και επ' αυτού. Την 6302 την ψηφίσαμε, κάναμε και τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Υπήρχε όμως και ένα σχόλιο, μια παρατήρηση συνδεδεμένη με αυτή την τροπολογία, την οποία όμως δεν την ψηφίσαμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε γι' αυτό τώρα. Α, κυρία Γκέντς, ναι. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι δεν ψηφίσαμε για το κείμενο αυτό καθεαυτό, για τα ε, μικροδάνεια, μικροπιστώσεις. Ό, ψηφίσαμε την τροπολογία για το νούμερο, αν θέλετε, λέει η Πρόεδρος. Τώρα το σχόλιο, την παρατήρηση, αν θέλετε, το κείμενο. Ψηφίζουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τροποποίηση του σχολείου, του, στην 6302. Για το 6302 υπερψηφίσαμε την αλλαγή του αριθμού. Ψηφίσατε όλοι. Contre. 3 contre et 2 pour. Αυτοί που δεν μπορούν να ψηφίσουν, 3 ε, κατά και 2 υπέρ. Πέρας της ψηφοφορίας. 41 votants. Ψήφισαν 41, 24 υπέρ, 10 κατά και 10 αποχές. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Σρότερ που μας ε, υπέδειξε το λάθος. Προχωρούμε τώρα στην ε, γνωμοδότηση. Παράγραφος 1. Τροπολογία 2 του εισηγητή. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Τροπολογία 3. Ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Τροπολογία της κυρίας Φιγκερέιδο. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 5. Φιγκερέιδο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 6 της Φιγκερέιδο, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 9, προφορική τροπολογία του κυρίου Καμπρνός. Υπάρχει αντίρρηση, αντίθεση για την προφορική αυτή προ... τροπολογία. Είστε κατά Οπότε δεν την ψηφίζουμε εφόσον υπάρχει κάποιος κατά. Προχωρούμε στην προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπάρχει κανείς αντίθετος. Κύριε εισηγητά έχετε το λόγο. Αποσύρεται η προφορική τροπολογία. Πολύ ωραία τροπολογία 7 της κυρίας Φιγκερέιδο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μετά την παράγραφο 10, τροπολογία 8 της κυρίας Γκιόνης. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 του κυρίου Χιούζ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την παράγραφο 18, τροπολογία 10 της κυρίας Φικηρέιδο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προχωρούμε τώρα στην τροπολογία 11 Guns Hughes και προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπάρχει αντίθεση για την προφορική τροπολογία. Όχι. Ωραία λοιπόν. Τροπολογία 11 τροποποιημένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 19 τροπολογία 12 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την αιτιολογική σκέψη σε τροπολογία 1 της κυρίας Φιγκερέδο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πείτε μου εσείς δεν έχετε κάρτες τι ψηφίζετε. Donc je rajoute deux voix pour. δύο υπέρ, ψήφους υπέρ. πέρα της ψηφοφορίας. Σαράντα ψηφίσαντες, υπέρ, 0 κατά 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Αν όλε οι ψηφοφορίε ε, γίνονται έτσι, τότε θα είμαστε η πιο αρμονική επιτροπή. Προχωρώ τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξη, που είναι το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Έχουμε τρεις υποθέσεις και θέλω να τις εξετάσουμε ξεχωριστά. Αυτό σας προτείνω. Μία υπόθεση... Η υπόθεση της Ισπανίας από την Καταλωνία και της Πορτογαλίας για κάποιε επιχειρήσει που βρίσκονται στο βορρά και στο κέντρο της χώρας. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, ήθελε ήδη από χτέ ε, να αποφανθεί για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Η επιστολή που απεστάλλει μετά από γραπτή διαβούλευση και με τους συντονιστές ε, και με τα μέλη της Επιτροπής Εργασίας σας έχει διανεμηθεί. Αυτή η επιστολή επιβεβαιώνει τα αιτήματα της Πορτογαλίας και της Ισπανίας για αυτές τις δύο υποθέσεις που συνδέονται με τη βιομηχανία, με την κλωστοϊφαντουργία ε, και που οδήγησαν σε διάφορες παρατηρήσεις και σχόλια και από πλευρά συντονιστών και από πλευρά ομάδας εργασίας Παρόλα αυτά δεν απερίφθησαν ε, τα αιτήματα των δύο αυτών χωρών. Περί τίνος πρόκειται, ποιες παρατηρήσεις ε, έγιναν. Ε, φέρουν επί της φύσης των διοικητικών δαπανών και κάποιων άλλων γενικόλογων θεμάτων, αλλά τίποτα, καμία λεπτομέρεια. Τώρα, υπάρχει το αίτημα της Γερμανίας στα πλαίσια της υπόθεσης Νόκια, τα μέλη της ομάδας εργασίας που συνεδρίασαν προχθές ε, θέλησαν να αναθεωρήσουν το σχέδιο ε, της επιστολής και θέλουν να επανασυνεδριάσουν πριν να σταλεί στα μέλη της Επιτροπής ε, το, η επιστολή. Θα ήθελα να σας θυμίσω τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναθεώρηση του σχεδίου και να προτείνω στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 29 Σεπτεμβρίου να συζητήσουμε επί της ουσίας το θέμα και να συζητήσουμε και την ίδια την επιστολή. Να την εγκρίνουμε ε, κατόπιν ή να την απορρίψουμε. Προέκυψε λοιπόν ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου επιστολής. Υπάρχει μια σειρά ε, στοιχείων που ήδη είναι γνωστά. Πρώτον, πώς ε, ε, τα, οι διοικητικές ε, δαπάνες εντοπίζονται. Ποια, πόσο λεπτομερής μπορεί να είναι η εικόνα που μπορούμε να έχουμε για τις διοικητικές δαπάνες. Για αυτό το θέμα προς το παρόν εκρεμεί η ουσιαστική απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν, για τον κατάλογο των δικαιούχων των κονδυλίων που θα κινητοποιηθούν μέσα στο Ταμείο έχουμε ερωτηματικά για την επικάλυψη που υπάρχει ανάμεσα στα κονδύλια που διανέμονται από το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και αφετέρου τα κονδύλια από το Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ η απάντηση που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας οδηγεί να αποταθούμε στη γερμανική κυβέρνηση για σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κινητοποίηση των κονδυλίων και στα δύο ταμεία και να ζητήσουμε διόρθωση των ε, χρονοδιαγραμμάτων που έχει παρουσιάσει. Τέλος, άλλη πολύ σημαντική ερώτηση είναι αν υπάρχει δυνατότητα να ε, κινητοποιήσουμε το Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το ταμείο σε περιπτώσεις όπου οι εργαζόμενοι δεν ε, εποφελούνται άμεσα από κάποια κατάρτιση ή κάποια ε, παροχή για την ανακύκλωσή τους, για την επανακατάρτισή τους. Ε, φαίνεται ότι σε αυτή την περίπτωση ικανοποιεί τα μέλη της ομάδας εργασίας η απάντηση που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε εργαζόμενος που λαμβάνει βοήθεια από το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει δικαιούται μάλλον μία ενίσχυση για την κατάρτιση ή την επανακατάρτιση χωρίς να χρειάζεται άμεσα να χρηματοδοτείται αυτή η δράση κατάρτιση από το ίδιο το ταμείο, μπορεί να προέρχονται τα κονδύλια και από άλλα ταμεία, έστω και εθνικά. Θελήσαμε να εμπλουτίσουμε τι ανταλλαγέ μα στην Επιτροπή, εστιάζοντα προσοχή μα σε δύο σημεία βασικά. Πρώτον, η ΑΠΕ η ευαισθησίας για το θέμα των φύλων που υπάρχει στον κανονισμό έχει επίσημο χαρακτήρα κατά τη γνώμη μας. Ε, αν κρίνουμε από την εξέταση και τη συνέχεια που δίνεται στους φακέλους, αφενός ε, και αφετέρου ε, τα μέλη της ομάδας εργασίας θέλουν να υπάρχει μια σαφέστερη εικόνα σε σχέση με το Πώ συνδέεται το Ταμείο προσαρμογή ε, στην παγκοσμιοποίηση με άλλε εθνικές ενώσει, οι οποίες όμως δεν έχουν προσδιοριστεί, δεν έχουν οριστεί ποιε είναι προς το παρόν σαφώ. Αυτά είναι τα σημεία που θέλω να εγείρω. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που έγιναν. Στο παρόν στάδιο δεν καλούμαστε να αποφασίσουμε για την υπόθεση Νόκια και το αίτημα της Γερμανίας, αλλά μπορούμε να ακούσουμε τους ε, συναδέλφους μας για να εμπλουτίσουμε τις ε, συζητήσεις ε, της ομάδας εργασίας. Ο κύριος Γιωβίν έχει ζητήσει το λόγο, με ενημερώνει η γραμματεία. Όχι, όχι, δεν το ζήτησα για αυτό το λόγο. Απλά ήθελα να ζητήσω από την Πρόεδρο να μην ε, σπέβδει τόσο πολύ όταν ψηφίζουμε, διότι δεν προλαβαίνουμε να παρακολουθήσουμε τον κατάλογο της ε, ψηφοφορίας ε, και ξέρετε θέλουμε τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε όταν χρειάζεται αυτό και... Αφήστε που έχετε τυπώσει με πολύ μικρά γράμματα αυτό τον κατάλογο της ψηφοφορίας και δυσκολεύομαι να την παρακαλουθήσω. Και με τη διερμηνία ε, υπάρχει μια, ακόμη μια μικρή καθυστέρηση και ορισμένες φορές δεν προλαβαίνουμε το, το χέρι να σηκώσουμε για να ζητήσουμε το λόγο γιατί πάει πάρα πολύ γρήγορα η ψηφοφορία. Ε, σας παρακαλούμε λίγο πιο αργή, λίγο πιο, λίγο πιο ήρεμα να γίνεται η ψηφοφορία γιατί ορισμένες φορές ε, μιλάμε για σημαντικά ζητήματα και το πόρισμα, το τελικό πόρισμα των εργασιών μας είναι η ίδια η ψηφοφορία μας δημιουργεί πρόβλημα το να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε με τόσο ταχύς ρυθμούς. Μάλιστα, είναι ένα θέμα που δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα. Θα μάθουμε να συμβιώνουμε, θα μάθουμε να προσαρμόσουμε τους ρυθμούς μας. Όλοι τελικά μαθαίνουν να ψηφίζουν γρήγορα, ξέρετε, για να ε, εξοικονομούμε χρόνο για την ουσιαστική συζήτηση. Αλλά λαμβάνω φυσικά υπόψη αυτά που μας είπατε. Η κυρία Ελιζαμπέτ Μογά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Για την ε, κοινή μας ε, δουλειά για αυτά τα δύο θέματα θέλω να σας πω τα εξής. Ε, δεδομένη συζήτηση που έχουμε κάνει, χτες συγκεκριμένα που κάναμε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, Βλέπω με χαρά σήμερα ότι μπορώ να υποστηρίξω ε, αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε για το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας για τις περιπτώσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ε, και δεδομένων των απαντήσεων ε, που πήραμε, και σχετικά με το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα της ισότητας των φύλων, Με χαρά δηλώνουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε την υποστήριξή μας γιατί για την κλωστοϊφαντουργία είναι εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Υπάρχουν περιοχές ε, επλήγησαν από μαζικότητα τις απολύσεις ε, και ε, μιλάμε για 1.600-1.700 εργαζομένους αυτές τις μαζικές απολύσεις προκύπτει ε, σαφώς ότι πρέπει να είναι δικαιούχος κάθε εργαζόμενος αυτών των παροχών του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και κατά περίπτωση πρέπει να εξετάζεται η παροχή βοήθειας ε, και ε, πρέπει να προσφέρεται μία εξατομικευμένη κατάρτιση για κάθε έναν από αυτούς τους εργαζόμενους. Για την υπόθεση Νόκια, ε, συμφωνώ μαζί σας και προσθέτω ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στα, για τα περιφερειακά ταμεία. Εσείς μιλήσατε για τα εθνικά ταμεία. Εγώ σας μιλώ και προσθέτω ότι πρέπει να επικρατεί διαφάνεια και για τα περιφερειακά ε, ταμεία, η Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε. Γιατί πέρα από το ΕΚΤ και το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν και άλλα ταμεία που μπορούν να επικουρήσουν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και χρειαζόμαστε την συζήτηση. Ε, κυρία, ο κύριος Σέρκας και η κυρία Φιγκυρέιντου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνεχίζω στην ίδια άγουσα με την κυρία Μωρά για να πω ότι καταρχάς σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες και την τόσο αποδοτική και γρήγορη εργασία η οποία μας επιτρέπει να ε, φτάσουμε στην πηγή του προβλήματος στις ε, περιοχές λοιπόν οι οποίες πλήχθησαν από την παγκοσμιοποίηση ε, κυρίως σε ένα τομέα ο οποίος είναι τόσο ευάλωτος όπως είναι η κλωστοϊφαντουργία. Ε, στην περιοχή της Καταλωνίας υπάρχουν χιλιάδες άτομα τα οποία πλήττονται. Ε, πλέον ε, σήμερα κοιτούν προς την Ευρώπη με περισσότερη ελπίδα. Δεν θεωρούν ότι είμαστε... Ε, ε, κουφή στα προβλήματά τους, κοφεύουμε όταν ε, μας τα αναφέρουν. Ευχαριστώ λοιπόν ε, την ομάδα εργασίας και το γεγονός ότι τα εξετάζεται κατά περίπτωση. Τώρα για την περίπτωση της Γερμανίας νομίζω ότι είναι ε, υψή να είμαστε το ίδιο γρήγοροι, το ίδιο αποτελεσματικοί και να εξετάσουμε ε, πολύ επισταμένα τα ευρωπαϊκά ταμεία ώστε να μην εξαντληθούν για το μέλλον. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν πολύ επισταμένα και θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή οδό. Όταν υπάρχουν διάφορε περιπτώσει, ε, θα πρέπει την κάθε μία να την εξετάζουμε στην ουσία τη και να μην περιμένουμε να λυθούν όλες ε, διαμιάς. Να λαμβάνουμε τις ε, οι οποίε θα είναι σοβαρέ, αλλά τα ταυτόχρονα θα έρχονται και αρκετά γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φιγκυρέντο και και η κυρία Ντανίτα Ζασλοβιέκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη ε, γιατί ήδη οι συνάδελφοι έκαναν ε, πολλές παρατηρήσεις. Θα ήθελα Αναφερόμενοι στην ομάδα εργασίας και για την, ε, να ευχαριστήσω για την υποστήριξη ε, που μας εδόθη και για το θέμα της Πορτογαλίας και για το θέμα της Ισπανίας ε, γιατί έχουν βυθιστεί στην ανεργία οι εργαζόμενοι και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να κινηθούμε ταχαίως ε, για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Η αίτηση ήδη έχει υποβληθεί από το 2008 τώρα για την υπόθεση Nokia. Δεν θα ε, αποφανθώ για αυτό το ζήτημα επί της αρχής το υποστηρίζω, αλλά πρέπει να εμβαθύνουμε στη συζήτηση. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Κυρία Ζαζοφιέσκα δεν θέλει το λόγο, οπότε ο κύριος ε, Τόμας Μάνε είναι ο τελευταίος εγγεγραμμένος ομιλητής. Ε, <clears throat> Eigentlich müsste ich Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ως Γερμανός βουλευτή ίσως δεν θα έπρεπε να μιλήσω για τη Γερμανία. Ίσως θα έπρεπε να μιλήσω για την Ισπανία, για την Πορτογαλία και από εκεί και πέρα τη Γερμανία την αφήσω απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, ε, παρόλα αυτά θα πω μερικά πράγματα για την Nokia, για τον τομέα της κινητής ε, τηλεφωνίας. Ε, η, τι έγινε, έκλεισε το εργοστάσιο του Μπόχουμ και η, ανεργία στην Γερμανία αυτή τη στιγμή ε, στην περιοχή του Μπόχουμ είναι ευτυχώς και λέω ευτυχώς 7% πρέπει βέβαια να μειωτηθεί περαιτέρω αλλά τι να κάνουμε λοιπόν ε, είδα τη παρουσίαση πάντως της περίπτωση της ε, γερμανικής ε, περίπτωσης θεωρώ ότι παρουσιάζεται πολύ λεπτομερώς και σωστά το θέμα συμφωνώ με την Ισπανία και την Πορτογαλία για το ε, για το το, κείμενο αλλά Τώρα μιλάμε μοναχά για την Νόκια. μην ξεχνάμε την Όπελ. Η Όπελ έρχεται, είναι πρώτον πυλών και δεν θα αφορά μοναχά το Χάν στο Χέσεν, την περιοχή που προέρχομαι εγώ, αλλά θα αφορά και άλλους. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μπάστος και η κυρία Ούτε Στάινμπρουκ θέλουν να πάρουν τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Συγχαίρω την ομάδα εργασίας για την απόφαση στην οποία κατέληξε στα αιτήματα αυτά, κυρίως για το πορτογαλικό αίτημα. Η κατάσταση στην Πορτογαλία οφείλεται στην πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, κυρίως στην ε, βόρεια ε, περιοχή της Πορτογαλίας, διότι η περιοχή αυτή είναι εξαρτώμενη από την κλωστό εφαντουργία και αυτό και πλήχθηκε από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ε, Παγκοσμιοποίηση ε, μπορεί να βοηθήσει τέτοιες περιοχές όπως είναι αυτή η Πορτογαλική, οι οποίες ε, πλήχθηκαν από τις αρνητικές συνέπειες του ανταγωνισμού των σημαντικών προϊόντων από χώρες ε, που είναι αναδυόμενες οικονομίες, όπως για παράδειγμα η Κίνα. Χάρη λοιπόν στο Ταμείο οι αρνητικές επιπτώσεις έχουν μετριαστεί σε σημαντικό βαθμό. Η χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση θα μπορέσει να συγκρατήσει και τις αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση. Όταν παρουσιάστηκε το αίτημα, όπως ε, πολύ σωστά υπόθηκε, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ σοβαρή, αλλά δεν ήταν τόσο δραματική όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι στο εγγύς μέλλον το, το Ταμείο Προσαρμογής ε, για την Πιαγκοσμιοποίηση, που όπως γνωρίζουμε είναι ένα ταμείο το οποίο ε, το έχουμε εμπνευστεί ε, με βάση την αρχή της αλληλεγγύης θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσει να αποτελέσει και την κατάλληλη απάντηση σε καταστάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν και στη χώρα μου αλλά και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούτα Στάινρουκ και στη συνέχεια η Συντόνια Γένσκα. Äh, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ε, την ανάγκη να υποστηριχθεί όχι γραφειοκρατικά εν πάση περιπτώσει αλλά πολύ γρήγορα η υπόθεση της Νόκια οι εργαζόμενοι εκεί ήδη έχουν πληγεί χάσαν τη δουλειά τους θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια και στήριξη πάρα πολύ σύντομα θα πρέπει να βοηθηθούν να ενταχθούν και πάλι στην αγορά εργασίας γι' αυτό σας παρακαλώ γρήγορη προώθηση και υποστήριξη Ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος, κυρία Συντόνια Ζέψκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία πρόεδρε. Ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα ήθελα να σας πω ότι και η Επιτροπή Προϋπολογισμών συζήτησε το θέμα αυτό εχθές και εκεί υποστηρίζονται αυτές οι προτάσεις Η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα για μένα, διότι κατανοώ λίγο και πώς έχει το υπόβαθρο σε αυτές τις ε, περιπτώσεις, σε αυτές τις αιτήσει. Και με λυπεί το γεγονός ότι ελάχιστες από αυτές τις αιτήσει ε, φτάνουν από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα ετήσιο ε, όριο 500 εκατομμυρίων ευρώ και εμείς έχουμε δαπανίσει μόνο 5 εκατομμύρια φέτος νομίζω. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να στέλνουν περισσότερες αιτήσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόνο 3-4 χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της κρίσης. Θα πρέπει να υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Επομένω, ε, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν περισσότερες αιτήσει και θα υπάρχουν και περισσότεροι που θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτή τη στήριξη και ε, σαφώς ε, και η Επιτροπή προπολογισμών, αλλά και η δική μα η Επιτροπή ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να κάνει τη δουλειά τους και να ενημερώνει τους πολίτε για την ύπαρξη αυτού του ταμείου. Ε, γιατί και το είπα και εγώ στην αρχή της παρέμβασής μου για την Ισπανική και την Πορτογαλική υπόθεση ε, είχαμε υπενθυμίσει αν θέλετε στις, στην Επιτροπή Προπολογισμών την ε, δική μας θέση Ε, στάλει μια επιστολή στο συνάδελφό μας κύριο Λαμασούρ τώρα για τη γερμανική υπόθεση θα ξανακουβεντιάσουμε το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 29 Σεπτεμβρίου θα δούμε και την επιστολή και θα ψηφίσουμε τώρα γενικό, γενικότερα για το ταμείο αυτό νομίζω ότι θα ξέρετε ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός που διέπει το ταμείο αυτό για να μπορεί το ταμείο να κινητοποιείται με χαμηλότερα κατόφλια κινητοποίηση αν θέλετε ε, και έχουμε ένα κατόφλι πεντακοσίων εργαζομένων τώρα που απολύονται Επίση, επίσης ε, η συμμετοχή του Ταμείου ανέρχεται στο 75% του κόστους και όχι στο 50% που ήταν πριν. Θέλω να πω ότι οι αλλαγές αυτές που έγιναν τώρα στο Ταμείο διευκολύνουν ουσιαστικά τη χρήση του Ταμείου αυτού και Πιστεύω ότι θα κινητοποιηθεί και θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο στο μέλλον του Ταμείου για αυτούς που δυστυχώς το έχουν ανάγκη. Αυτά. Κυρίες και κύριοι για σήμερα προχωρώ στο επόμενο και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. συγγνώμη, ο κύριος Τόμας Κυρία Πρόεδρε, δείτε, ίσως πρέπει να το θέσουμε το θέμα ως διαδικαστικό. Ε, στο παρελθόν ε, έχουμε πει επανειλημμένως ότι δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις γιατί θα πρέπει να αναφερόμαστε σε γενικότερα θέματα κτλ. Λοιπόν, ωραία. Εδώ όμως ε, στην περίπτωση του Ταμείου ε, Παγκοσμιοποίησης δεν θα πρέπει να ε, κρατήσουμε αν θέλετε αυτή τη στάση ούτως ή άλλως εδώ πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα πράγματα θέλουμε τα πράγματα αυτά να τα μάθει και το κοινό γι' αυτό λοιπόν να μην τα κουκλώσουμε όπως το παρελθόν γιατί ε, δεν αλλάζουμε στάση Πρόεδρος, εδώ έχουμε πρόβλημα διότι όλη η ιστορία της κινητοποίησης του Ταμείου δεν είναι να κάνουμε θεωρητικές συζητήσεις αλλά πολύ πρακτικά να σε και γρήγορα να κάνουμε πράγματα τους ώστε να στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από την παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία και προσπαθούμε ε, και εμείς να ε, προσαρμοστούμε για να είμαστε, να είμαστε όμως και αποτελεσματικοί συγχρόνως. Τώρα τη συζήτηση στην οποία αναφερθήκατε θα μπορέ, τη συζήτηση αυτή θα πρέπει να την κάνουμε όταν θα συζητήσουμε την ετήσια έκθεση του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση. Τον Ιούλιο ε, θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση αυτή για το 2008. Ξέρω ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ετοιμάζεται να κάνει και αυτή η σχόλια. Λοιπόν, τότε όταν θα κουβεντιάζουμε την ετήσια έκθεση θα ε, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις συζητήσεις αυτές. Η κυρία Μωράν ζητεί το λόγο. Ποιος άλλος? Η κυρία Ντελή και μετά κλείνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Μωρά, μετά από την παρατήρηση του Τόμας Μαν θα ήθελα να πω το εξή. Συνειδητοποιούμε ότι για να είμαστε σωστοί και να πρέπει να επαγρυπνούμε για σχετικά με την, το πώς εξελίσσονται τα αιτήματα που υποβάλλονται για το ταμείο αυτό. Πώς πάει η κατάσταση. Τροποποιήθηκε στην αρχή της χρονιάς όντως ο κανονισμός του ταμείου. Αλλά αρκεί η τροποποίηση αυτή. Έχουμε την οικονομική κρίση. Από πράγματα πρακτικά δηλαδή στην καθημερινότητα. Άρα είναι απαραίτητο να κάνουμε τις συζητήσεις αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Ντελή. Ντελή θα ήθελα να μου πείτε τι περιθώρια, περιθώρια ευελιξίες υπάρχουν, τι μπορεί να γίνει για την περίπτωση της Νόκια. Φύγανε από τη Γερμανία, πήγανε στην Νοτιοανατολική Ασία. Ε, υπάρχουν κυρώσεις, πρόεδρος. Η ομάδα εργασίας και με το θέμα αυτό. Δείτε, Εμεί εδώ καλούμεθα να πούμε κατά πόσο πρέπει να κινητοποιηθεί το Ταμείο ή όχι. Το Ταμείο κινητοποιείται υπέρ των εργαζομένων και όχι υπέρ των επιχειρήσεων. Η Νόκια έκανε απολύσεις. Συζητήθηκε το πώς έγιναν οι απολύσεις αυτές. Η πλειοψηφία της ομάδας εργασίας ε, θεώρησε ότι η μέθοδος με την οποία έγιναν διάφορες απολύσεις δεν επηρεάζει το κατά πώς θα κινητοποιηθεί ή όχι το ταμείο και τη βοήθεια που θα δοθεί στους εργαζόμενους. Τώρα εσύ θέτε το θέμα των κυρώσεων ε, λόγω λόγο της μετά επίση του εργοστασίου από την Ευρώπη στο εξωτερικό και τα και τα Αυτά όντως είναι θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Εμείς εδώ όμως τους μιλούμε για το ταμείο που κινητοποιείται υπέρ των εργαζομένων και αυτό το αίτημα το η ομάδα εργασίας το συζήτησε και είπε ότι βεβαίως δεν πρόκειται να, κυρώ, να επιβληθούν κυρώσεις στους εργαζόμενους που χάσαν τη δουλειά τους. Το άλλο είναι μια γενικότερη συζήτηση, πρέπει να γίνει αλλού. Αυτά για το σημείο αυτό κυρίες και κύριοι. Προχωρούμε σε ένα, στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που σχετίζεται με ναι. μια μεγάλη συζήτηση που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει για τις πολιτικές προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής θητείας. Η Επιτροπή μας έχει κάποιες ευθύνες ή κάποιες αρμοδιότητες. Τι θα κάνει Επιπλέον θα έχουμε μια καινούργια κομισιόν σε λίγο. Πώς θα αντιδράσει η Επιτροπή μας. Βεβαίως 60% των μελών αυτής της Επιτροπής είναι νέα μέλη. Ε. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε βλέποντας τα θέματα τα οποία μας έχουν κληροδοτηθεί από τους προκατόχους μας, ένα αυτό, τι εκρεμεί λοιπόν. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να χαράξουμε μια στρατηγική που θέλει να ακολουθήσει η Επιτροπή μας. Λοιπόν, για τα... για το τι μας κληροδότησαν μετά από την χτεσινή και τη σημερινή συνεδρίαση ε, μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποια θέματα που είναι μπλοκαρισμένα και τα λέω τώρα λίγο ανάκατα πρώτον το θέμα είναι η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων συμπληρωματικής σύνταξης από το 2007 έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο το θέμα αυτό. Η Επιτροπή θέλει να ξαναξεκινήσει τη συζήτηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φτιάξει και μια πράσινη βίβλο. Οπότε θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Οι υπηρεσίες κοινοφελείς, υπηρεσίες, ε, υπηρεσίες κοινοφελούς συμφέροντος. Είναι ε, πολύ... Αυτές οι υπηρεσίες αποκλείονται από την ίδια την οδηγία των υπηρεσιών. Και αντί να αναλυφθεί πρωτοβουλία εδώ για το θέμα αυτό όπως μας είχε πει η Επιτροπή έγινε μονάχα μια ανακοίνωση σχετικά. Τρίτο θέμα που, μπλοκα... που έχει μπλοκαριστεί είναι το θέμα του χρόνου εργασίας. Είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει για τη, την διαδικασία που θα εφαρμοστεί ενάντια σε εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία αυτή του χρόνου εργασίας. Η Τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις στην αρχή της χρονιάς. Τελικά μπλοκαρίστηκε μεταξύ των επιτρόπων το θέμα αυτό. Άλλο θέμα το οποίο εκκρεμεί το Ευρωπαϊκό έτος 2010 ε, κατά της ε, ένδυας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να κάνουμε σχετικά, να αξιολογήσουμε, να δούμε τι πολιτικές υπάρχουν σχετικά και αν υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις ε, που μπορούν να εκτελεστούν στο μέλλον και αν υπάρχει κάτι στο νομοθετικό πρόγραμμα της Κομισιόν στην επόμενη την επόμενη ίσω κομισιόν. Λοιπόν, τώρα το επόμενο θέμα βεβαίω είναι το, η έκθεση της κυρίας Μπάουερ, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, δεν θα τα ξαναπώ αυτά. Μιλάμε για, τους, για τις κινητές δραστηριότητες στο μέτρο μεταφορών. Δεν λέω τίποτα άλλο. Μετά έχουμε τα, τη μικροχρηματοδότηση, μικροδάνεια, μικροπιστώσεις κτλ. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίασή μας. Ε, εν τω μεταξύ έχουν κατατεθεί α, τροπολογίες για τη δημιουργία μιας νέας γραμμής, μιας νέας θέσης στον προϋπολογισμό ε, για τα, τις μικροπιστώσεις. Άλλα θέματα τώρα καινούρια που θα πρέπει να πραγματευτούμε είναι αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας που βεβαίως δεν αφορά μοναχά τη δική μας την Επιτροπή, είναι γενικότερο θέμα και μετά η οδηγία για του εποχιακούς εργαζόμενους των ναι, υπηκών τρίτων χωρών γιατί η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση προετοιμάζει ένα σχέδιο οδηγίας για το θέμα αυτό. Ωραία προσθέτω μεταξύ των θεμάτων που ίσως θα πρέπει να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό που ακούσαμε σήμερα το πρωί της απόσπασης των εργαζομένων επίκαιρο και καυτό θέμα αυτό και υπάρχουν και άλλα βέβαια θέματα στην μελέτη που είδαμε χτες ε, υπάρχουν πολλά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν φαντάζομαι. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ περαιτέρω. Ε, παραμένω εδώ. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα και παλιά και καινούργια που πρέπει να δούμε. Επίσης θέλω να πω δύο πράγματα. Πέρα από τις βασι, τη βασική δουλειά που πρέπει να κάνει η Επιτροπή μας υπάρχουν και άλλα πράγματα πρέπει να εντάξουμε στην καθημερινή μας δουλειά. Ίσως θα πρέπει να δούμε πώς η πολιτική απασχόληση εντάσσεται ή συναρθρώνεται με άλλες πολιτικές, με την οικονομική πολιτική παραδείγματος χάρη, άλλες πολιτικές ε, εκπαίδευση κλπ. Η στρατηγική της Λισαβόνας και η συνθήκη της Λισαβόνας βεβαίω ε, περιμένουμε να εγκριθεί κλπ. Αλλά ε, βιώνουμε και μια οικονομική κρίση. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, υπό αυτές, λόγω όλων αυτών των πραγμάτων να κάνουμε και κάποιες σκέψεις για το πώς συναρθρώνεται η πολιτική απασχόληση με άλλες πολιτικές ή πώς θα έπρεπε να συναρθρώνεται. Και κάτι τι άλλο ε, για την καινούργια θητεία είναι ένα θέμα που έμεσα αναφέρθηκε στην περασμένη θητεία μέσω της έκθεσης Richard Witt, Howitt, για τις επιχειρήσεις. Λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διατρέχουμε και επειδή πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια καινούργια αρχή Ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθούν και οι μισθοί και η συμμετοχή των εργαζομένων στα διοικητικά και άλλα συμβούλια των επιχειρήσεων ε, για το πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να επηρεάσουν περαιτέρω το τι κάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτά όλα βέβαια προ... Προ... προϋποθέτουν συνεργασία και με άλλες ε, επιτροπές οικονομικών και τα λοιπά, βιομηχανίας. Α, ε, το λέω αυτό για να πω ότι θα ήθελα στην επόμενη θητεία η επιτροπή μας να είναι παρούσα, παρούσα. Ε, και ελπίζω να μην μακρηγόρησα υπερβολικά θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα σε εκπροσώπους από διάφορες πολιτικές ομάδες για να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση στρατηγικής αν θέλετε που πρέπει νομίζω να κάνουμε για το μέλλον της Επιτροπής μας. Ξεκινούμε από τον κύριο Τσαμπαωρή και μετά με το λόγο στον κύριο Σέρκας. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα, κυρίως για την τελευταία φράση που είπατε. Έχω κάποιες δυσκολίες επί της ε, διαδικασίας. Εμένα θα με χαροποιούσε ιδιαίτερα αν υπήρχαν κάποια έγγραφα, ένα γραπτό κείμενο το οποίο θα συνοψίζει ε, τα πράγματα βάσει και το οποίο θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ξέρουμε βέβαια πολύ καλά ποια είναι τα θέματα τα οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, είναι εξελίξη, μπορούμε να καθορίσουμε και τι προτεραιότητες έχουμε που θα μπορούσαν να αφορούν είτε κάποιες ε, γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας, εκθέσεις πρωτοβουλίας είτε άλλα έγγραφα, αλλά κατά την άποψή μου θα ήταν καλύτερο αν ε, θεωρήσουμε αυτή τη συζήτηση ε, ως μια διαδικασία ενημέρωσης, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να ξέρουν ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, αλλήλων και να μπορούμε να συζητήσουμε επί τη βάση ενός ε, συγκεκριμένου, πιο διαρθρωμένου κειμένου. Μεταξύ των προτεραιοτήτων μας είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλάβουμε και το θέμα των ατόμων με αναπηρία, διότι πρόκειται για άτομα τα οποία είναι τα πιο ευάλωτα δεδομένης και της κρίσης. Επαναλαμβάνω λοιπόν, και εμείς θα σκεφτούμε εις βάθος ε, ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, και στα πλαίσια της πολιτικής μας ομάδας και εάν μας δοθεί και ένα γραπτό κείμενο θα είναι ίσως καλύτερο να ε, συζητήσουμε πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος, διότι ίσως ε, αυτό που είπε ο κύριος ορί, το να έχουμε δηλαδή κάποιο μικρό κείμενο θα μας ήταν χρήσιμο ε, ήδη υπάρχει. Μας το έχουν ε, ετοιμάσει η γραμματεία, εξαιρετική δουλειά και πραγματικά είναι λίγο ε, μια ιστορική αναδρομή της Επιτροπής και ε, στον καθένα δίνονται και λίγο οι προσανατολισμοί για το μέλλον. και επομένως ε, μπορούμε να συζητήσουμε ίσως άμα έχουμε και ένα έγγραφο όπως είπε και ο κύριος Σωρή ε, που θα μας δίνει και λίγο κάποιους πολιτικούς προσανατολισμούς και κάποια πράγματα ε, για το τι μέλη γενέστε. Και εμείς ως πολιτική ομάδα, ως σοσιαλιστές ε, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει. Μας ενδιαφέρει και λίγο το ε, περιβάλλον της θητείας σας αυτής. Ε, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον αρκετά κρίσιμο και λόγω της οικονομικής και της κοινωνικής κατάστασης, αλλά και γιατί μόλις βιώσαμε και κάποιες εκλογές οι οποίες για άλλη μια φορά μας κατέδειξαν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, ακούν από το κοινοβούλιο ε, μία γλώσσα που δεν είναι πάντα κατανοητή και υπάρχει και ολοένα μειούμενο ενδιαφέρον το οποίο διαπιστώνουμε κυρίως μεταξύ των εργοζομένων και τις ε, πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, ανεξάρτητα ιδεολογίας, ξέρουν πάρα πολύ ότι ε, το ευρωπαϊκό ε, πολύ καλά ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ε, έχει και μια κοινωνική συνιστόσα. έχουμε όμως μια κρίση και εμείς η στρατηγική μας ως σοσιαλιστές είναι να έχουμε μια κάποια πρόοδο η οποία θα είναι οριζόντια και θα είναι συνολική για όλους. Να έχουμε μια ατζέντα η οποία μπορεί να μην αντικατοπτρίζει το 100% των ανησυχιών μας αλλά να είναι ένα βήμα προς τα μπρος σε αυτό το οικοδόμημα και να δημιουργήσουμε μια νέα κοινωνική ατζέντα για την Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι από αυτό προκύπτουν ακριβώς δύο στοιχεία. Το από τη μια έχουμε την οικονομική κρίση και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στους πολίτες τη σαφή εικόνα ότι υπάρχει μια αυθεντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να καταπολεμήσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της, κοινωνική, της οικονομικής κρίσης, κυρίως για την ανεργία, κυρίως για να δοθούν νέες δυνατότητες στους εργαζομένους που χάνουν τις θέσεις ε, απασχόλησής τους και ε, η Ευρώπη δεν είναι μόνο ένας χώρος συζήτησης, είναι ένας χώρος στον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις και αναζητούνται λύσεις για την οικονομική κρίση και στην κοινωνική της διάσταση και δεν συζητάμε μόνο τον κόσμο των επιχειρήσεων. Εντάξει, οι επιχειρήσεις είναι η λύση των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά υπάρχουν άνδρες και γυναίκες που πάσχουν και εμείς όπως είδατε και σήμερα το πρωί με τη συζήτησή μας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση ότι κάτι υπάρχει. Αυτό είναι το ένα πλαίσιο. Και το άλλο πλαίσιο είναι ότι δεν έχουμε αρκετά μέσα. Μα το είπαν και οι Σουηδοί Υπουργοί σήμερα το πρωί. Έχουμε πολύ λίγα οικονομικά μέσα, πολύ λίγα πολιτικά μέσα και Δεδομένου ότι θα έρθει και η νέα συνθήκη της Λισαβόνας και η νέα στρατηγική της Λισαβόνας, ίσως να είναι η κατάλληλη στιγμή. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Έτος ε, για την Ένδια και, την, ε, και το Κοινωνικό Αποκλεισμό το 2010. Ίσως ήγηκε η ώρα λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το νομικό πλαίσιο για τους ε, ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευάλωτοι, που είναι ανάπηροι, που είναι ασθενείς, ε, που είναι νέοι, που είναι ηλικιωμένοι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει μια σειρά από συγκεκριμένε πρωτοβουλίες. Εσείς ε, είπατε ότι πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την οδηγία για τον ε, χρόνο εργασία. Αυτή είναι μια οδηγία η οποία ουσιαστικά έχει γίνει το σύμβολο, το λάβαρο για την ε, ε, σχέση που πρέπει να έχουμε με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε και με ένα θέμα που αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο οικονομική ατζέντα η ατζέντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι και μια κοινωνική ατζέντα και θα πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ευελιξία μεν για τι επιχειρήσει, αλλά και την ασφάλεια για του εργαζομένου δεν θα πρέπει να είναι μόνο η ευελιξία, θα πρέπει να είναι μια ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινάσει ε, άλλους εννέα ναι, μήνες διαλόγου με τους ε, κοινωνικούς εταίρους. Μακάρι να καταλήξουμε σε αποτέλεσμα με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά τελικά θα βρεθούμε στο Σεπτέμβριο και μπορεί να ε, βρεθούμε πάλι να συζητάμε την ίδια οδηγία. Ελπίζω να μην φτάσει γιατί οι κοινωνικοί εταίροι θα μας όσουν δώσει μια λύση. Ευχαριστούμε κυρία Μαρκίνη, συντονίστρια των φιλελευθέρων δεν είναι εδώ, οπότε θα δώσω το λόγο στην ε, κυρία Λίν. Ευχαριστώ. Ναι, ε, ήδη ακούγονται πολλά ενδιαφέροντα σχόλια. Στην τωρινή θητεία θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την υλοποίηση. Τα τελευταία δέκα χρόνια που είμαι εγώ εδώ στο Κοινοβούλιο δεν έχουμε ασχοληθεί με τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Εγώ θα ήθελα να αυξήσουμε το ρόλο μας, ε, τον ελεγκτικό μας ε, ρόλο προς την εφαρμογή. Όπως είπε και ο κύριος Σόρη, καλό θα ήταν να εκπονηθεί ένα έγγραφο αν δούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, αν δούμε γιατί δεν έχει υλοποιηθεί σωστά στα διάφορα κράτη-μέλη και να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να διευκολύνουμε την εφαρμογή. Αυτό είναι μια καλή λύση και διάφορες άλλες επιτροπές εξετάζουν ακριβώς το ίδιο ζήτημα αλλά μου φαίνεται παράλογο. Συνέχεια προσθέτουμε νομοθεσίες ενώ δεν λειτουργούν αυτές που ήδη υπάρχουν ίσως να χρειαστεί να καταργηθούν κάποιες νομοθεσίες και αν ξαναχρειαστούν, εντάξει, ας ε, τις ε, παρεκπονήσουμε. Αλλά τουλάχιστον φροντίσουμε να εφαρμόζονται ε, σωστά τα, οι νομικές πράξεις κλειδιά για να μπορούν να συμμετάσχουν και να χρησιμοποιούν την νομοθεσία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάρη. Κάτι άλλο τώρα όπως ε, ε, σε σχέση με αυτό που έκανα με τον Στίφεν Χιούσε για τις τραυματισμούς από τις βελόνες, ενοχληθήκαμε και οι δύο γιατί περάσαμε όλη αυτή τη βαριά νομοθετική διαδικασία και ξαφνικά η κοινωνική εταιρεία είπαν όχι, θέλουμε να αποφασίσουμε εμείς. Παρ' όλα αυτά το καλοκαίρι ελήφθη απόφαση και ίσως θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, μεριμνήσουμε ώστε να δώσει τουλάχιστον συνέχεια σε αυτή την πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων. Βλέπω γνέφη και ο Στίφεν. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και ε, ε, κάτι άλλο είναι κατάργηση διακριτική μεταχείρισης ε, τώρα που έχουμε και τη Σουηδική Προεδρία. Αυτή τη φορά θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση προ το Συμβούλιο, ούτω ώστε ε, ε, μετά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στη δική μα Επιτροπή και μέσα από τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία, να φροντίσουμε ώστε να προκύψει μια συγκεκριμένη οδηγία. Ίσως να συνεργαστούμε καλύτερα με την, οδηγία πολιτικών με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών συγγνώμη, για να συγκεντρώσουμε τις δυνάμει μας και να πιέσουμε το Συμβούλιο. Αυτά προς το παρόν. Καλό είναι αυτό που είπε ο κ. Σόρη για ένα νέο έγγραφο και τα νέα μέλη τη Επιτροπής καλό θα ήταν να ε, έχουν ε, υπόψη ότι μπορούν να συνεισφέρουν στη διαδικασία γιατί υπάρχουν αρκετά νέα μέλη. Μπορούν να συμμετάσχουν λοιπόν ενεργά για τα επόμενα πέντε χρόνια. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους η κυρία Τζιν Λάμπερτ και κατόπιν ε, θα ακούσουμε τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ε, και η κυρία Μπάουερ θα πάρει πρώτη το λόγο. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε μαζί σας για την ανάγκη η Επιτροπής μας να είναι πανταχού παρούσα σε πολλές ε, από τις σημαντικές συζητήσεις οι οποίες είναι εξελίξει. Μία από αυτές, όπως μας είπατε κι εσείς, είναι η αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνα και να έχουμε μια νέα στρατηγική. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα συνδεθεί και με πολλά θέματα που σχετίζονται με τις συζητήσεις ε, που θα γίνουν στην Κοπενχάγη αργότερα για τις κλιματικές αλλαγές και την ε, ε, οικονομία η οποία θα έχει χαμηλή κατανάλωση άνθρακα και με τις επιχειρήσεις. Γίνονται πολλές εργασίες με τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων που ασχολούνται με οικολογικές θέσεις εργασίας, οικολογική απασχόληση και δεν έχουμε συνδεθεί καταλήλως με αυτό, με σοβαρό τρόπο τουλάχιστον μέχρι τώρα στην Επιτροπή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική διάσταση για μας, διότι δεν είναι μόνο θέμα του να έχουν θέσεις απασχόλησης οι ε, άνθρωποι, αλλά και τι τύπο απασχόλησης έσους ε, και τι συνθήκες εργασίας επικρατούν. Και ε, επίσης θα πρέπει να δούμε λίγο πώς μπορούμε να, να τη συνεχίσουμε αυτή τη μελέτη, διότι σχετίζεται και με τη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, και αν θέλουμε να έχουμε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους και να υπάρχει και κράτος δικαίου, θα πρέπει να δούμε, όπως είδαμε και από τη χθεσινή παρουσίαση, ε, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και τα δύο στοιχεία, και την ανάπτυξη και την αυτοαπασχόληση και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν και αυτές τις νέες μορφές, μάλλον όχι νέες μορφές, τις ε, διάφορες ποικιλομορφίε ε, εργασίας που έχουμε πλέον και αυτά μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να διασυνδέσουμε όλα αυτά τα υπόλοιπα στοιχεία με την αναθεώρηση στρατηγικής ε, ε, της Λισαβόνας και το πρόβλημα, πρόγραμμα ανάκτηση. Και επίση θα πρέπει να δούμε και τι σημαίνει αυτό με τις ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και το πρόγραμμα εργασία. Υπήρχε και ένα ερώτημα για την απασχόληση των νέων, όπως επίσης και την απασχόληση των ηλικιμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία. Πώς μπορούν όλα αυτά να συγκεραστούν, διότι βλέπουμε ότι γίνονται λίγα στην Επιτροπή μας ε, και δεν λαμβάνονται υπόψη και τα εθνικά προγράμματα δράσης. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που είπατε για την εφαρμογή, αν και νομίζω ότι μάλλον την εννοούμε διαφορετικά την εφαρμογή και τι θεωρούμε όλοι ως εφαρμογή, αλλά αυτό έχει σχέση και με τα θέματα που αφορούν ε, στις αποσπάσεις των εργαζομένων, ακόμα και για την, ε, ε, τους μεταφερόμενους εργαζόμενους που ακούσαμε χθε. Έχουμε μόνο 10% ελέγχους στους υπαλλήλους οδηγούς. Γιατί γίνεται αυτό, είναι θέμα νομοθεσίας ή έχει να κάνει με την εφαρμογή στα κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν να κάνουν κάτι. Ακούσαμε ότι έχουμε άτυπη εργασία, δήλωτη εργασία κλπ. εδώ στην Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε όλους αυτούς τους τομείς, κυρίως ε, για την ε, αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, και θεωρώ ως δεδομένο ότι μας ενδιαφέρει ως πολιτική ομάδα και το όλο θέμα της ε, ένδυας και της κοινωνικής ένταξης. Ευχαριστούμε. Πάμε στο δεύτερο στάδιο, στη συζήτηση. Δηλαδή, και θα ακούσουμε την κυρία Μπάουερ και την κυρία Μοχά. Κυρία Μπάουερ, πιστεύω ότι όλοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και διαβλέπουμε όλα τα προβλήματα που πρέπει να ρυθμιστούν πάρα αυτά. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που πρέπει να ρυθμίσουμε μέσα στην αγορά εργασίας μεταξύ αυτών των προβλημάτων. Υπάρχουν πολλά που μας επηρεάζουν, μας αφορούν άμεσα. Ε, στην Επιτροπή μας μιλάμε για τις δημογραφικές τάσεις και τα προβλήματα λόγω των νέων δημογραφικών τάσεων συγκεκριμένα. Και ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε πως η Επιτροπή μας θα έπρεπε να ασχοληθεί εντατικότερα με τα δημογραφικά προβλήματα. Ε, όμως θα έπρεπε να εκπονήσουμε ένα συγκεκριμένο έγγραφο για την γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Πιστεύετε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα και πρέπει να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Ε, κοιτάξτε, θα σας απαντήσω στο τέλος, αφού ακούσουμε και τις συναδέλφους. Η κυρία Μογά έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα... Ε, εμείνω σε τρία σημεία όπως και οι προηγούμενοι ομιλητές, όπως ο παραδείγματος χαρή ο κύριος Σέρκας. Στα πλαίσια της κρίσης αναθεωρείται το θεματολόγιο της Λισαβόνας. Υπάρχουν τρία όμως σημεία που δεν μπορούμε να παραλείψουμε. Πρώτον, εξυγχρονισμό του κοινωνικού διαλόγου. Σε μία περίοδο κρίσης πρέπει από νομοθετικής ε, πλευράς να φροντίσουμε να εξυγχρονιστεί ο κοινωνικός ε, διάλογος, ε, διότι συχνά διαπιστώνουμε ελλείψεις οι οποίες δημιουργούν, έχουν καταστρεφικές συνέπειες στην αγορά εργασίας. Αυτή την περίοδο της κρίσης πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με την ευθύνη που πρέπει να φέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μεγάλοι όμιλοι ε, επιχειρήσεων σε σχέση ε, με το κλείσιμο κάπου ποιον υπεργολάβων. Γιατί ξέρετε, το 90% της δουλειάς των υπεργολάβων προέρχεται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, και ποια η ευθύνη για την ανεργία, ποια σχέση υπάρχει ε, με την, ε, πώς θα επιμερίσουμε την ευθύνη ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους υπεργολάβους. Είχαμε πολλές σοβαρές περιπτώσεις, κυρίως στη Γαλλία, και πρέπει οπωσδήποτε να εσκύψουμε στο θέμα της εταιρική ευθύνης. Κάτι άλλο τώρα, πάλι στα πλαίσια της κρίσης, Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή πώς να αναβαθμίσουμε τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους ε, οι μισθωτοί για να προσαρμοστούν στις νέες θέσεις εργασίας ή να ε, ενταχθούν στη νέα αγορά εργασίας, ε, πώς κυρώνουν την, και πιστοποιούν τα προσόντα τους και την εμπειρία τους. Ε, ήδη ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, αλλά ε, στην πράξη δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Δεν είναι αποτελεσματικό ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το θέμα. Και το ίδιο ισχύει και με τα συστήματα κατάρτισης ε, και θα ήταν εξαιρετικά επικερδές να λειτουργούμε και λίγο πιο δραστήρια, λίγο πιο προληπτικά στον τομέα αυτό. Η κυρία Σαρία Σαγιά και ο κύριος Στίφεν Χιούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάφοροι συνάδελφοι είπαν ήδη ότι τα επόμενα χρόνια θα χαρακτηριστούν σε μεγάλο βαθμό από την τωρινή κρίση. Ε, όσο επιδεινώνεται η κατάσταση, τόσο υποφέρουν ε, αυτοί που βρίσκονται σε, στις πιο, οι πιο ευπαθείς ε, πληθυσμιακές ε, ομάδες και συγκεκριμένα οι πιο ευπαθείς ομάδες της αγοράς εργασίας, δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες, παραδείγματος χάρη, η μακροχρόνια άνεργη. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για μαζική ανεργία των νέων και αυτό θα οδηγεί σε μαζικό κοινωνικό αποκλεισμό όλη η ζωή κάποιου ατόμου μπορεί να καταστραφεί ε, ε, εξαιτία αυτού και παραμένει ανεκμετάλλευτο το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό μας προβληματίζει και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στον τομέα της ε, παιδείας. Επίσης, η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είχαμε ακρόαση εχθές Ακούσαμε και συναδέλφους από το Κογκρέσο τον ΗΠΑ που ε, μας μίλησαν για αυτό το ζήτημα. Πρέπει οπωσδήποτε στην Ευρώπη να αποφύγουμε δύο παράλληλες ε, αγορές εργασίας, ε, μία επίσημη και μία γκρίζα γιατί αυτό θα οδηγήσει και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και φυσικά σε ε, υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε ο κύριος ε, Στέφεν Χιούζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα γιατί πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τις σκέψεις μας εν ώψη της ακρόασης με τον επόμενο Επίτροπο ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Πρέπει να ενημερωθούμε για τα ζητήματα ότως ώστε να θέσουμε σωστές ερωτήσεις ε, στον υποψήφιο Επίτροπο για να καταφέρουμε ήδη από τώρα να μας δώσει εγγυήσεις για, ε, για ολόκληρη τη θητεία του ή Πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη ακρόαση. Ε, έχω διάφορα σημεία. Ζητώ συγγνώμη να επαναλάβω κάτι που είπαν ήδη οι συνάδελφοι. Ένα επίγον πρόβλημα που πρέπει να ρυθμίσουμε ε, στα πλαίσια της κρίσης που αντιμετωπίζουμε ε, είναι ε, ο κόδωνας κινδύνου που κρούν αυτοί που ασχολούνται με τα δημοσιονομικά. Δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν παίρνουν κονδύλια από το ΕΚΤΕ, δεν απορροφούν ε, κονδύλια, δεν ζητάνε άμεσες πληρωμές από το ΕΚΤΕ. 30 με 40% των κονδυλίων του ΕΚΤΕ δεν θα απορροφηθούν και δεν θα δαπανηθούν επί τόπου παρότι εσχάτως απλουστεύσαμε τον κανονισμό. Δεν ξέρω τι δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω που κολλάει ε, το, το πράγμα. πρέπει να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως είναι το πρόβλημα οι αυστηρότατοι έλεγχοι. Πρέπει να τους καλέσουμε εδώ και να συζητήσουμε με τους εκπρόσωπου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς θα εφαρμόσουμε στην πράξη τον κανονισμό, τον απλουστευμένο κανονισμό για να απορροφηθούν τα κονδύλια. Ε, όπως είπατε Πρόεδρε, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για τις κοινοφελείς υπηρεσίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέκαθεν μας έλεγε ότι είναι δύσκολο να εκπονήσουμε τέτοιο έγγραφο εμείς ε, ζητήσαμε από δικηγόρους να συντάξουν μια οδηγία, αυτό το κάναμε πριν από δύο χρόνια και ε, τη δώσαμε την οδηγία, το σχέδιο οδηγίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τίποτα δεν έχει γίνει έκτοτε. Αυτό είναι το σύμβολο ε, της κατάρρευσης του κοινωνικού και εκτιμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν προσέξουμε. Έχει συμβολική αξία, πρέπει να μην το παρατήσουμε αυτό το θέμα η επισφαλή θέση εργασία, η ευελιξασφάλεια που ε, μας απασχόλησε ε, στην προηγούμενη θητεία αυτό ε, θα οδηγήσει επισφαλείς συνθήκες διαβίωση για όλο ένα και μεγαλύτερο αριθμό προσώπων. Έχουμε την μερική απασχόληση στην εξωτερική ανάθεση, διάφορες μορφές άτυπη εργασίας, τέτοια φαινόμενα είναι ενδυμικά σε χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να ρυθμίσουμε την κατάσταση και κυρίω νέοι ε, βρίσκονται σε τέτοιες επισφαλείς καταστάσεις, ε, δηλαδή όσοι φοιτούν ε, αναγκάζονται δωρεάν να δουλεύουν 4-5 χρόνια πριν καταφέρουν να βρουν μία δουλειά. Πρέπει να δούμε τους κανονισμούς, να μην επιτρέψουμε αυτή την εκμετάλλευση των νέων και αναφερθήκαμε πολλά στη, στην οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Μην ξεχνάτε ότι η απόφαση Λουξεμβούργου και Λαβάλ άνοιξε άλλο ευρύ φάσμα ερωτήσεων, ε, ανισορροπία ανάμεσα στι οικονομικέ ελευθερίε τη συνθήκη και ε, των θεμελιωδών ε, ελευθεριών έχουμε ένα σύνολο προβλημάτων που δημιουργούν αυτές οι αποφάσεις ε, του ΔΕΚ και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ε, δύσκολη. Έχουμε και δύο σχέδια ε, κοινωνικής δράσης, παραδείγματος χάρη για τις συλλογικέ συμβάσεις. Το ξέχασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι γίνεται, πρέπει να το δούμε και αυτό. Ε, με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές και τα λοιπά που γίνονται λόγω της κρίσης. Ε, πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα για να δούμε από πλευρά Ένωσης ποια πρότυπα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διατηρηθούν στην αγορά εργασίας, να παραμείνουν στην αγορά εργασίας ε, οι άνθρωποι και να μην γίνουν μακροχρόνια άνεργοι και να απομακρυνθούν από την αγορά εργασίας. Επίσης, ενημέρωση και διαβούλευση, όπως είπε σωστά η κυρία Μογάν, πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον κοινωνικό διάλογο για τις διαβουλεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Ε, και έχουμε τη σύμβαση για τον υπεράριθμο προσωπικό. Διάφορες οδηγίες που έχουμε από το 70, 70 ε, συγγνώμη, ε, και υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί για την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Ούτε καν καταφέρνουμε να ορίσουμε τι εστί διαβούλευση. ακόμη και στα πλαίσια των επιχειρησιακών συμβουλίων για τη διαβούλευση ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζομένους για την εταιρική ευθύνη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπατε για τους τραυματισμούς από τις βελόνες ε, τώρα έρχομαι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πούνε πότε θα μετατρέψουν σε οδηγία τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά δεν ξέρω αν έχει ε, ακόμη προσδιοριστεί η ημερομηνία τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ ευχαριστώ κυρία μετά το πολλά πράγματα ακούστηκαν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να προσθέσω μερικά ακόμη σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής έγινε λόγος για την οικονομική κρίση την οποία διατρέχουμε αυτή τη στιγμή και η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον και θα μετατραπεί από οικονομική σε κοινωνική κρίση υπάρχουν πολλοί ευάλωτες πολλές ευάλωτες ομάδες ε, πιο ευάλωτες από άλλες. Ο κ. Σωρή μας μίλησε για τα άτομα με α, αναπηρίες. Εγώ θα σας αναφέρω τους ΡΟΜ και έχουμε φτιάξει και μια έκθεση για τους Ρώμα. Η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και δύσκολη και ξέρουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη η πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα που θίγεται από την κρίση, από, τις, ε, από την άνηση μεταχείριση κτλ. είναι η Ρώμα θα πρέπει να υπάρχει κοινοτική πολιτική για τους Ρώμα. Πρόκειται για, σε τελευταία ανάλυση για 12 εκατομμύρια άτομα, μα λάβουμε υπόψη μας όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται μια μειονότητα αρκετά μεγάλη και μεταξύ των Ρώμα ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν και παιδιά, ε Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι ακόμη πιο ευάλωτα για εκτός από τον πληθυσμό των Ρώμ βεβαίως ευάλωτα είναι τα παιδιά την κοινωνία μας γενικότερα. Λοιπόν, θα πρέπει να φροντίσουμε τα παιδιά, τα παιδιά που ζουν σε φτωχές οικογένειες για να μπορέσουν να βγουν από τη φτώχεια, από την ε, ε δυστυχή κατάσταση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και όπως ακούστηκε ήδη ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με το κοινωνικό ταμείο Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τόμας Μάνι πρόεδρος Πρόεδρε ε, μια σύντομη παρατήρηση θέλω να κάνω και δύο σχόλια. Πρώτη παρατηρήση και σε σχέση με αυτά που είπε ο Στίβεν Χιούς. Βεβαίω θα ήταν πολύ σημαντικό να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες του κοινωνικού ταμείου. Παρόλα αυτά το κοινωνικό ταμείο είναι 50 ετών και το ταμείο αυτό λειτουργεί καλά και τα, τα, κονδύλια τα οποία διαθέτει το κοινωνικό ταμείο τελικά πάνε στη βάση, πάνε σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, δεν χάνονται σε κάποια μαύρη τρύπα στα διάφορα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να γελιόμαστε, το κοινωνικό ταμείο είναι επιτυχές. Τώρα έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Μπάουερ για τις ε, ε γενιές και κυρία Πρόεδρε, θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να δούμε τι γίνεται με τις τους ηλικιωμένους ή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα στην αγορά εργασίας. Ίσως θα πρέπει να διευρύνουμε και το τι εννοούμε στα δουλειά που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί. Ε, οι άνθρωποι θα τους συνδυάσουμε την εκπαίδευση, να συνδυάσουμε, τις, να φτιάχνουμε ομάδες πολλα, με μέλη από πολλές γενιές τους ώστε οι μεν να ε, βοηθούν με την πείρα τους τους δε και λοιπά και λοιπά. Και τέλος να πω και κάτι άλλο. Η κυρία Μέρκελ είπε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα διεθνές μοντέλο της αγοράς, εργα... της, ε, αγοράς ε, της οικονομίας αγοράς με κοινωνικό πρόσωπο, τη social market, αυτό που λέμε στη Γερμανία, για ούτως ώστε να μπορέσουν και άλλοι να χρησιμοποιήσουν αυτό το α, ε, διεθνές μοντέλο. Δεν ε, διαφημίζω τώρα την... Α, καγκελάριό μας απλώς λέω ότι πραγματικά πρέπει να φροντίσουμε μετά από τα αυτά που λέγαμε χτες για flexicurity και αυτά που βλέπουμε ε, τι γίνονται και στις διάφορες επιχειρήσεις και στα διάφορα κράτη-μέλη θα πρέπει πράγματι να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει τελικά το μοντέλο αυτό στην Ευρώπη, στη Γερμανία χρησιμοποιείται, απλώς θέλει μια καινούργια παρουσίαση για να τα ακολουθήσουν κι άλλοι. Η κυρία Γιακονσάρη παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, Περβάνς, διότι ξεκίνησες αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω η Γραμματεία να μπορέσει να εξορίξει κάποια διαμάντια από αυτή τη συζήτηση να ευχαριστήσω, ε, να, συγγνώμη, να σου εκφράσω τον χειρότερο μου φόβο. Με ανησυχεί ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο αυτή η παγκόσμια κρίση επηρεάζει την Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα κλείσουμε την πόρτα στη μετανάστευση και αν περιορίσουμε τη μετανάστευση σημαίνει ότι θα δώσουμε το πράσινο φως για την παράνομη μετανάστευση. Και η παράνομη μετανάστευση θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση των εργαζομένων με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Πιστεύω λοιπόν ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει να παραμείνει συνεχώς εν γνώση ε, των όσων συμβαίνουν στη σκιά της ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων. Εχθές κάποιος ε, μίλησε για την ελεύθερη μετακίνηση και είπε ότι ε, ουσιαστικά ο κόσμος υποχρεώνεται να μεταφερθεί από τη μία πλευρά στην άλλη. Ε, είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν εκεί που ε, έχουν μια θέση εργασίας και ορισμένες φορές απελάβνονται και τους στέλνουν πίσω στη χώρα τους. Μ' ανησυχεί ιδιαίτερα λοιπόν το σύγχρονο δουλεμπόριο Νομίζω ότι μια μέρα θα βρεθεί η γενιά μας ενώπιον του ε, Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη Χάγη γιατί κλείσαμε τα μάτια μας ε, ε, στην ε, νόμιμη μετανάστευση και ξεχάσαμε τι σημαίνει σύγχρονο δουλεμπόριο. Το σύγχρονο δουλεμπόριο σήμερα είναι χειρότερο από το δουλεμπόριο του παρελθόντος. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου παρατήρηση αν περιορίσουμε την μετανάστευση, αν έχουμε περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές, ε, θα έχουμε ε, πρόβλημα με την παράνομη μετανάστευση. Τώρα, έχουμε την πράσινη οικονομική ανάπτυξη. Τι μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προάγουμε την πράσινη ανάπτυξη. Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε τους νέους ανθρώπους για την ε, ε, ενεργειακή απόδοση. Αυτή είναι ερώτηση. Τρίτη παρατήρηση. Η Επιτροπή μας έχει πάλι μια σειρά από εκθέσεις. Το ίδιο και το Κοινοβούλιο. Την Άνοιξη εγκρίναμε την έκθεση Λέχτινεν Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε, διότι έχει να κάνει με την ε, γκρίζα οικονομία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον ορισμένες φορές να δείτε τι εκθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν και να δουν τι, συνέβη και να εξάγετε συμπεράσματα ως προς την αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριο Σέργιο Κομφεράτη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι οι εργασίες της Επιτροπής μας θα πρέπει να συνδέονται στενά με την πορεία της κρίσης. Η Ευρώπη κατελήφθη εξαπίνης, είχε υποτιμήσει τις πρώτες ενδείξεις οι οποίες σαφέστατα καταδείκνυαν τι συνέβαινε σε άλλες χώρες, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, και κατά συνέπεια αυτή τη στιγμή πληρώνει σε όλες τις χώρες ε, βαρύτατα αυτή την καθυστέρηση, την οποία δεν μπορούμε και να ανακτήσουμε. Ορισμένες φορές λοιπόν... Ε, ε, δεν υπάρχουν και εμπειρίες να μας δείξουν τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί αυτά είναι όλα καινοφανή και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Διότι τους μήνες που μας περιμένουν, αν συνοδεύονται μία, από μια περαιτέρω πτώση του εισοδήματος ε, ή των θέσεων εργασίας ε, για άντρες και γυναίκες, σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε ένα καθεστώς πανικού. Και αυτό φυσικά θα έχει συνέπειες και στη συμπεριφορά των ανθρώπων, τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά. Και επίσης υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο. Θα πρέπει τώρα να σκεφτούμε πώς μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε τη διέξοδα από την κρίση όταν θα υπάρξει. Ε, πέρα από τους χρονικούς περιορισμούς, αν δεν έχουμε στεναρό προσανατολισμό και των πολιτικών και των ε, θεσμικών οργάνων, υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθούν μοντέλα τα οποία θα οδηγήσουν στην παλιά ε, ευρωπαϊκή κουλτούρα. Αντί, για παράδειγμα, να θεωρηθεί ευκαιρία το περιβάλλον, θα θεωρηθεί τσάκος απορριμμάτων για να έχουμε κάποια αντιγωνιστική θέση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν θα έχουμε σε καμία περίπτωση την πράσινη οικονομία που ευελπιστούμε να έχουμε. Πιστεύω ότι κάποια θέματα, τα θέματα των δικαιωμάτων, ε, θα μπορούσαν να δουν τα κατόφλια τους να πέφτουν για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε κάποια στοιχεία και μπορεί να, μην, να χαθεί εκεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να το ανανεώσουμε, αλλά για να το ανανεώσουμε θα πρέπει να έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Παραδείγματο χάρη, η σχέση μεταξύ κοινωνικών εταίρων είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την κοινωνική σχέση αυτή και θα πρέπει να έχουμε και οποιαδήποτε θετική ένδειξη μπορούμε, θετική εξέλιξη μεταξύ ανθρώπων που εκπροσωπούν το χώρο της εργασίας και το χώρο των επιχειρήσεων. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να ενισχύσουμε τα στοιχεία της κοινωνικής προστασίας, διότι όπου υπάρχει συνοχή, υπάρχουν και οι προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και για να ε, ε, δώσουμε μια νέα όθηση στην οικονομία. Η κοινωνική συνοχή είναι ένα από τα πιο βασικά, πιο σημαντικά στοιχεία της ε, ανταγωνιστικότητας. Δεν ε, μας εκπλήσει το γεγονός ότι ο Μπάρακ Ομπάμα συζητά ε, το θέμα της υγειονομικής περίθαλψης των ατόμων και δεν σκέφτεται μόνο τους ανθρώπους, σκέφτεται και την αξία που θα έχει η συνοχή από εκεί και πέρα στον ε, κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσουμε και ένα διάλογο με τον τομέα των επιχειρήσεων για το θέμα της ε, κοινωνικής ευθύνης. Η Ευρώπη το έθεσε το θέμα αυτό σε ανύποπτο χρόνο. Το να επανέλθουμε λοιπόν να το συζητήσουμε τώρα μπορεί να είναι χρήσιμο και για το παρόν αλλά και για τις μελλοντικέ μας προοπτικές. Ευχαριστούμε κύριο και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω πως είναι πολύ χρήσιμη η συζήτηση που κάνουμε. Είναι πολύ θετικό που κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα και θα ακούσουμε και ακούμε ενδιαφέρουσες απόψεις. Αλλά δεν έχει κανένα πλαίσιο η συζήτησή μας. Δεν λέω ότι είναι άχρηστη η συζήτηση, αλλά χρειαζόμαστε κάτι γραπτό σε πέντε χρόνια δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, όλα τα προβλήματα του κόσμου. Χρειαζόμαστε ένα κατάλογο, να καταγράψουμε ποια προβλήματα που πρέπει να ρυθμίσουμε. Η κρίση είναι ύψιστη προτεραιότητα, κατόπιν έχουμε παγκόσμιου χαρακτήρα προκλήσεις, έχουμε τη δημογραφική πρόκληση, τα συνταξιοδοτικά συστήματα, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν κατά προτεραιότητα. Έχουν γίνει αλλαγές ε, στα συνταξιωτικά και τα ασφαλιστικά συστήματα σε όλα τα κράτη. Και εφόσον μιλάμε για συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση, μην ξεχνάμε και το, τη διακρατική διάσταση του ζητήματος και προβλήματα ανεπίλητα στην Ευρώπη, προβλήματα που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο. Ε, μας μίλησαν πολύ για τις ε, άτυπες ε, μορφές εργασίας. Χτες μιλούσαμε για τους ψευδοαπασχολούμενους. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτές τις κατηγορίες των εργαζομένων. Η γραμματεία έχει ε, πάρει σημειώσεις και θα μπορούσε ίσως να συντάξει ένα έγγραφο με όλες τις προτεραιότητες, ούτω ώστε να είναι λίγο πιο εστιασμένη η συζήτησή μας ε, έτσι. Ε, θα ξέρουμε και ποιες ερωτήσεις θα θέσουμε στον υποψήφιο επίτροπο. Μιλώ γκρικά όπως θα έχετε παρατηρήσει, γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα και σε ένα άλλο κράτος μέλος, στη Σλοβακία, υπάρχουν υπάρχει, μια, ε, ε, υπάρχει απαγόρευση ομιλίας της Ουγγρικής σε κάποιους χώρους ε, εργασίας. Και ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το νέο νόμο που τους απαγορεύει να μιλάνε Ουγγρικά στη Σλοβακία. Θέλω να γίνει ευρέως γνωστό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, για αυτό το τελευταίο που είπατε δεν νομίζω ότι αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή μας και ότι πρέπει να το σημειώσει η Γραμματεία. Αλλά πάντω ενημερώσατε του συναδέλφου, Η κυρία καριμάτελη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τωρινή ε, οικονομική κρίση πλήττει τους πλέον αδύναμους, ε, του, τις πλέον ευαίσθητες ομάδες. Είπατε, Πρόεδρε, ότι υπάρχει το θέμα τη δημοκρατική συμμετοχή τη επιχειρήση. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει. Οι μισθωτή. πρέπει να, πρέπει να τη φωνή των μισθωτών σχετικά με την λειτουργία της ε, ε, επιχείρηση. Θέλω να μιλήσουμε για τις ανισότητες. Θα ζητήσει κανείς από τον Δηλαδή, ε, ποιο μισθωτό θα πει ότι είναι λογικό το αφεντικό του να κερδίζει 600 φορέ περισσότερα χρήματα από ότι αυτό. Οι ανισότητες λοιπόν, οι εισοδηματικές ανισότητες ε, πρέπει να μας απασχολήσουν και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων έχει συζητήσει ήδη το θέμα και ελπίζω και ε, να μας απασχολήσουν και εμάς σύντομα. Η συνάδελφός μου μας μίλησε για την Κοπενχάγη. Νομίζω ότι ε, μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε για αυτές τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, να συμφωνήσουμε και να κάνουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις. Τέλος, η υγεία στο χώρο εργασίας. Ακόμη υπάρχουν εργάτες ε, που εργάζονται σήμερα σε επικίνδυνα εργοστάσια. Δεν την χάνουν καμίας προστασίας. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τους προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει άλλος ομιλητή, ομιλητής, οπότε σας προτείνω εν είδη προσωρινού συμπεράσματος να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, ζήτησαν ε, συνάδελφοι ένα κείμενο. Ε, επίσημα να πούμε ποιες θα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες δηλαδή της Επιτροπής μας μέσα σε ένα έγγραφο. Ε, θα δούμε ποια θα είναι η μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί και πέρα κάθε πολιτική ομάδα θα αυτοπροσδιοριστεί, ας το πω έτσι, θα προσδιορίσει ε, τις προτεραιότητές της ε, σε σχέση με τη νέα Επιτροπή. Βέβαια, από κοινού εμείς θα κινηθούμε για να κάνουμε μία σύνοψη της ε, συζήτηση μάλλον για να τροφοδοτήσουμε τις ε, μελλοντικέ ε, συζητήσεις. Σχετικά με το κληροδότημά μας, σας παραπέμπω στο πακέτο καλωσορίσματος των νέων μελών που έχει βάλει στη διάθεσή σας η γραμματεία και εκεί αναφέρονται όλα αυτά τα σημεία κυρίως για, τα τρέχον, για τους τρέχοντες φακέλους, μελλοντικούς φακέλους, φακέλους της Επιτροπής μας και στις 29 Σεπτεμβρίου θα ζητήσω από τη Γραμματεία να πάρει να κάνει μία σύνοψη ε, της παρουσίασης ε, που έγινε ε, στα μέλη με το που αρχίσαμε τις εργασίες μας. Ο κύριος Μπουζίκ ζήτησε από τους Προέδρους των Επιτροπών ε, να ε, αποταθεί στον μελλοντικό πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων που δεν έχει ακόμη οριστεί, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα και να του δώσει μια επιστολή με τις ε, προγραμματικές ε, προτεραιότητες. Επί την βάση του κληροδοτήματος της προηγουμένης θητείας και της συζήτησης που μόλις κάναμε, θα είναι μια σύντομη επιστολή, αυτός είναι ο στόχος και θα υποδείξουμε απλά τι επιθυμεί η Επιτροπή μας. Η συζήτηση που κάναμε είναι πολύτιμη. Ε, θα φτιάξουμε ένα ερωτηματολόγιο εν ώψη της ε, ακρόασης ε, του ή της του μελλοντικού υποψηφίου, της μελλοντικής υποψηφίου για τη θέση του της Επιτρόπου. Και επί τη βάση της συζήτησης θα ζητήσω από τη Γραμματεία να προετοιμάσει ένα σχέδιο, ένα πρόχειρο για αυτό το ερωτηματολόγιο. Τέλος, στη συνεδρία των συντονιστών θα ε, ασχοληθούμε με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής. Θα δούμε ποιες, ε, θα προσδιορίσουμε για ποιες εκθέσεις πρωτοβουλίας, ιδίας πρωτοβουλίας θέλουμε να ζητήσουμε την έγκριση και ε, θα δούμε ποιες μελέτες θα μας ενδιέφεραν ε, να γίνουν. Αυτά τα τρία σημεία λοιπόν. Θα απαντήσουμε στον κύριο Μπούζα και θα στείλουμε την επιστολή. Θα φτιάξουμε το ερωτηματολόγιο για τη μελλοντική ακρόαση του υποψηφίου επιτρόπου και ε, θα εξετάσουμε το πρόγραμμα εργασιών με τους συντονιστές για να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τη σημερινή συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα θα αρχίσουν να διαγράφονται οι προτεραιότητες της ε, Επιτροπής, αλλά και των διαφόρων πολιτικών ομάδων στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Αυτά για σήμερα. Ε, ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση στις 29 Σεπτεμβρίου και σας λέω ήδη από τώρα ότι για τις 30 υπάρχει μια βεβαιότητα ε, σίγουρα θα συνεδριάσουμε όλη τη μέρα στις 29. Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη μπορούμε ή όχι να καταργήσουμε τη συνεδρία στις 30 γιατί στις 29 θα ε, έχουμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε και μία ακρόαση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τους Φακέλους που είναι δική μας ε,